Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω όλους ε, θερμά ε, και θα ήθελα να καλωσορίσω ε, κυρίες, κυρίως την Επίτροπό μας, την κυρία Κιονκίν, η οποία θα λάβει το λόγο ως πρώτη σήμερα το πρωί και κατόπιν θα είναι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Έχουμε στο χρόνο μας, στη διάθεσή μας μία ώρα χρόνο. ξεκινάμε λοιπόν, ελπίζω να είναι ευχάριστη η μέρα μας, έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Κυρία Κιονκίν, σας καλωσορίζουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα και σε άλλες συνεδριάσεις, ε, από την εντολή και ε, μετά, Εμεί θέλουμε να ασχοληθούμε με όλου του τομεί τη έρευνα. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου προσφέρετε ευκαιρία να συζητήσω μαζί σα το ε, 7ο πρόγραμμα, την ενδιάμεση αξιολόγηση ε, και ένα γενικότερο στρατηγικό πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία και τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα επίση να έχω ανταλλαγή απόψεων μαζί σα σε σχέση με την Πράσινη Βίβλο που ε, δημοσιεύτηκε πρόσφατα για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση του 7ου πλαίσιο, πλαίσιο. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για να υπάρχει μια αμερόληπτη άποψη, για να εντοπιστούν προβλήματα και για να αναζητηθούν και οι λύσει. Η αξιολόγηση έλαβε χώρα από μια ομάδα 10 ανεξάρτητων εμπειρογνώμων υπό τον Ρόλφ Άντεμπεργκ, ο οποίο είναι ο Γενικό Διευθυντή του Σουηδικού Ερευνητικού ε, Ινστιτούτου για Έρευνα και Ανάπτυξη. Ε, φαντάζομαι ότι τον γνωρίζετε πλέον ε, όλοι σας πολύ καλά μετά τη χθεσινή συζήτηση που από, από ό,τι άκουσα ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν λοιπόν συμπεράσματα στην αξιολόγηση εμπειρογνώμονες, περιορίζεται σε 10 συστάσεις για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 7ου προγράμματος και αναφέρουν και ορισμένες ιδέες για μελλοντικά προγράμματα. Οι αντιδράσεις των κρατών μελών και των άμεσα εμπλεκόμενων διαφορεμένων ήταν πολύ θετική. Αναφέρεται ότι η έκθεση αξιολόγηση έτυχε καλή αποδοχή ε, ω μια εμπεριστατωμένη άποψη για το πού ακριβώ βρισκόμαστε και πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Η δομή της απάντησης της Κομισιόν ε, δέχεται και τις 10 συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Η απάντηση περιλαμβάνει ε, τα απορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμών όσον αφορά τους στόχους και την εφαρμογή μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Ε, υπογραμμίζει επίσης ότι η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να στηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 συμπεριλαμβανομένων και των φιλόδοξων στόχων της πρωτοβουλίας Ναυαρχίδα όπω αποκαλείται. Επίσης, ε, ε, καλούνται οι υπόλοιποι οργανισμοί να αναπτύξουν και εκείνοι κοινέ προσεγγίσεις. Ένα παράδειγμα λοιπόν μιας προσέγγισης που απαιτεί την υποστήριξη όλων ε, των θεσμών είναι η ανάπτυξη και λήψη μέτρων για τη μελλοντική χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι οι προσπάθειες για να ενισχυθεί η ε, χρηματοδότηση ε, των ε, χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει απαντήσεις που έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2007. Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό και περίπλοκο θέμα, το οποίο αναφέρεται στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων, δηλαδή στο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής ορισμένων κρατών μελών. Το πρόγραμμα πλαίσιο αφορά την επιστημονική αριστεία και θα υπάρχουν πάντα χώρες οι οποίες είναι κάτω από το μέσο όρο. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ανησυχεί για το κατά πόσον ε, θα υπάρχει υποαποτελεσματικότητα και κατά πόσον υπάρχουν ε, δυνατότητες να υπάρξει ανάκαμψη. Τώρα, όσον αφορά την Υπό εκπροσώπηση, Η Κομισιόν καταρχήν θέλει να ακούσει ε, μέσα από τις ε, διαβουλεύσεις και έτσι θα, βοηθεί, θα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα πλαίσιο κοινή στρατηγικής για να διαπιστώσουμε πως είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερη συνεργασία με τα διευθυντικά ταμεία στην πρακτική. Και αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο των προτάσεων για την ε, χρηματοδότηση, εκ νέου χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Επίσης, θα έχουμε φόρα σε διάφορα επίπεδα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα θέματα και τα προσκόμματα και εκεί θα εξεταστούν λειτουργικά στοιχεία ε, διαχείρισης του προγράμματος όπως επίσης και διαρθρωτικά θέματα ε, στις ε, εμπλεκόμενες χώρες. Το να εντοπίσει κανείς την ευπή εξειδίκευση αυτό είναι καθοριστική σημασία. Όλες οι χώρες σε όλους τους τομείς πρέπει να αισθάνονται ότι εμπλέκονται και αν υπάρχουν συγκεκριμένοι φραγμοί αυτοί πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως αν τα προγράμματα χρηματοδότησης θέλουμε να συμβάλλουν στους στόχους της Ευρώπης 2020 με τη στήριξη της Παγκόσμιας δεν πρέπει να υπονομεύουμε την αρχή της αριστείας στη χρηματοδότηση καινοτόμων προγραμμάτων. Γιατί εμεί θέλουμε το καλύτερο. Το Συμβούλιο των Υπουργών κάλεσε την Επιτροπή να αναλύσει ποσοστά συμμετοχής ε, και στο τέλος του έτους να υπάρξει αναφορά να ε, υποβληθούν νέα μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις ε, προτινόμενες εξελίξεις η ουσία της ε, πράσινης βίβλου πρέπει να συγκριθεί με το παρελθόν και ως μια σημαντική δέσμευση ε, για την ε, εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επίσης ε, θα πρέπει τα προγράμματά μας ε, να εξορθολογιστούν, να ακολουθήσουν απλουστευμένες διαδικασίες και παράλληλα να διασφαλίσουν μια αμυγός ευρωπαϊκή προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι αυτή η στρατηγική προσέγγιση είναι μόνο μόνος δρόμος προς τα εμπρός εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξου στόχου του 2020. Και με χαρά άκουσα ότι η προσέγγιση αυτή συμβαδίζει με κάποιες συστάσεις στο σχέδιο έκθεσης κυρίας Μέρκης, ε, το οποίο σχέδιο θα ψηφιστεί στην επόμενη Ολομέλη του Μαΐου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο μέλλον αν θέλουμε να αναδυθούμε ισχυρότεροι από την οικονομική κρίση. Και μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να κινητοποιήσουμε επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Μόνο μέσα από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να οθήσουμε τους ερευνητές θέση να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργαστούν πέρα από τα σύνορα. Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, οργανώσει ε, σε όλη την Ευρώπη διαγωνισμούς ε, με επιδίωξη την αριστεία. Ως εκ τούτου η έρευνα και η κινητομία πρέπει ένα καθοριστικό στοιχείο ενός οξυντερκούς ε, κοινοτικού προπολογισμού και αυτό είναι καθοριστικό εάν πραγματικά θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 και της Ένωσης Καινοτομιών. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πιο ε, συνδυασμένο τρόπο. Θα βελτιώσει τους δεσμούς ανάμεσα στην κοινοτική χρηματοδότηση διαφόρων κρίκων της ε, αλυσίδα καινοτομιών όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίε που προσφέρονται στην αγορά. Επίση, θα διασφαλίσει ότι όλα τα στοιχεία της χρηματοδοτησή μα συμβάλλουν στο να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις που πλήττουν την Ευρώπη σε τομεί, όπω είναι η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια, η ασφάλεια των τροφίμων. Το πλέον σημαντικό είναι ότι θα επιτρέψουμε στην Ευρώπη αυτέ τι προκλήσει να τι μετατρέψει σε ευκαιρίε και να δημιουργήσει περισσότερη αύξηση και θέσει εργασία. Όλα αυτά θα ισχύουν για την παραδοσιακή έρευνα στα κλασικά προγράμματα πλαίσιο, αλλά και για τι νέε μεθόδου συνεργασία, όπω τώρα προωθούνται από, την, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Κοινοτομία και την Τεχνολογία. Επίση, θα ισχύουν για την κοινοτομία στι εταιρείε που αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την ανταγωνιστικότητα και το πλαίσιο για την κοινοτομία. Με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο σκοπεύουμε να παράσχουμε μια ευθυγραμμισμένη ε, προσέγγιση και μια σειρά μέτρων που θα καλύπτουν την εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα δημοσιονομικά μέσα για την έρευνα και την κοινοτομία αυτή τη στιγμή είναι διασκορπισμένα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και επίσης το πλαίσιο για την ε, τεχνολογία και την κοινοτομία. Εδώ υπάρχουν δάνεια από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο που τα δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. το πλαίσιο για την ε, έρευνα και την καινοτομία δίνει και δανειοληπτικές εγγυήσει και διευκολύνσεις ε, δανείων για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα διευθυντικά ταμεία επίση στηρίζουν μια σειρά από οικονομικά προγράμματα για τι δυνατότητε καινοτομία στι διάφορε επιμέρου περιοχέ. Το να ευθυγραμμιστούν όλα αυτά τα εργαλεία χρηματοδότηση είναι κάτι που θα έρθει να συμπέσει με την περίοδο επαναπρογραμματισμού του ευρωπαϊκού προπολογισμού και καλύτερη κατανομή και ισορροπία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε επιτυχημένοι στην ε, ευρωπαϊκή έρευνα και την καινοτομία και τον προπολογισμό τη, πρέπει να δείξουμε με μεγάλη σαφήνεια πώ κάνουμε τα πράγματα, πώ μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά όλα αυτά τα εργαλεία και πώ κάθε ευρώ που ξοδεύουμε δαπανάται σωστά. Έτσι θα έχουμε ριζοσπαστικέ αλλαγέ στον τρόπο που χρηματοδοτούμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Μέσω αυτή τη πράσινη βίβλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων, αναζητώντα τι απόψει των φορέων για το πώ θα επιτύχει όλα αυτά κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εύχομαι ότι βάσει τη πράσινη βίβλου θα μπορέσουμε να είμαστε δραστηριοί και να ενεργήσουμε άμεσα. Οι διαβουλεύσει θα τελειώσουν στι 20 Μαου και το αποτέλεσμα θα υποβληθεί για να συζητηθεί σε διάσκεψη τη Βρυξέλλε στι 10 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τι προτάσει τη για τη μελλοντική ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία και τα προγράμματά του πριν το τέλο τη φετινή χρονιά. Σε αυτό το πλαίσιο, η δική σας άποψη για την πράσινη βίβλο θα ε, συμβάλλει στην προετοιμασία μας των ερχόμενων αυτών προτάσεων. Ε, άκουσα ότι η κυρία Ματίας ως εισηγήτρια για την πράσινη βίβλο έχει ήδη διαμορφώσει μια άποψη και ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας λίγα λόγια για την ε, οικονομική διευκόλυνση, το εργαλείο διευκόλυνσης για την κατανομή του κινδύνου. Εδώ έγινε αξιολόγηση από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου η κυρία Ερίκα Μάνη, πρώην ε, βουλευτή, ε, προείδρευε και νομίζω ότι είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε μαζί του τον περασμένο Οκτώβριο. Ήταν θετική αξιολόγηση του οργάνου αυτού από του εμπειρογνώμονε. Από το 2011 ω το 2013 ζητάτε η άμεση απελευθέρωση των 500 εκατομμυρίων ε, ευρώ για την χρηματοδότηση του 7ου προγράμματος πλαισίου, της δεύτερης δηλαδή θέτας αυτής του προγράμματος, που είναι πολύ σημαντική για την συνέχεια λειτουργία του 7ου προγράμματος πλαισίου και για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις αιτήσει για δάνεια στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου για κοινοτομία και έρευνα. Έως το 2011, ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία έχει τύχει συμφωνίας ε, από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και μέχρι τώρα τα 250 εκατομμύρια ως το 2011 είχαν εγκριθεί. Ε, τώρα τα 500 εκατομμύρια προκειμένου να ταμιευθούν πρέπει να τύχουν τη έγκριση του Κοινοβουλίου. Εάν αυτό γίνει από πλευρά Κοινοβουλίου, νομίζω θα δώσουμε ένα πολύ θετικό μήνυμα προ την ε, κοινότητα των ερευνητών και επιστημόνων. Νομίζω ότι ο κύριο Οντί, που είναι υπεύθυνο για την έκθεση περί αξιολόγηση του 7 προγράμματο πλαισίου και οι σκιώδει εισηγητέ, συνεργάζονται για να καταλήξουν σε μια έκθεση με περιεχόμενο και υψηλή ποιότητα. Είναι πολύ σημαντική η δική σα τοποθέτηση σε σχέση με την δική μα πορεία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Κύριε Γκροστέτ, παρακαλώ, έχετε το λόγο πρώτη. μια στιγμή, διακόπτει ο Πρόεδρος. Να λάβουμε υπόψη μας ότι στις 10 ώρα θα σταματήσουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Γι' αυτό Ίσως δεν μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο. Έχουμε 8, 9 που έχουν στήσει το λόγο. Πρώτη κυρία Κροστέτ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για τις εξηγήσεις που μας έδωσε όσον αφορά την πράσινη βίβλο και τις ε, συζητήσεις που κάνετε. Για αυτό το πρόγραμμα, το ερευνητικό, εγώ θέλω να αφαιρθώ στη μεταφορά τεχνολογίας γιατί σήμερα όλο και περισσότερο βλέπουμε να μεταφέρεται τεχνολογία στις αναδιόμενες χώρες, χώρες οι οποίες δεν θα έπρεπε να θεωρούνται πια αναδυόμενες. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει αμοιβαιότητα, γιατί δεν είναι δυνατόν επαόριστο να θεωρούμε ότι η μεταφορά αυτή τεχνολογία θα γίνεται προς μία μόνο κατεύθυνση και ότι εμείς δεν θα μπορούμε να αποφελούμεθα από έρευνες που γίνονται σε αυτές τις χώρες. Εμείς θα θέλαμε οι σχέσεις μας να μην είναι μονόδρομος, να πάψουμε πια να θεωρούμε ότι η δικιά μας η βιομηχανική πολιτική είναι η τέλεια και να γνωρούμε άλλες ε, έρευνες που γίνονται στον κόσμο. Οι αναδυόμενες χώρες εξάλλου χαίρουν δημοσίων ενισχύσεων κατ' εξαίρεση με υπερβολικά ποσά που τους δίνουν την δυνατότητα να αγοράσουν τη δικιά μας την τεχνολογία ή να κερδίζουν διαγωνισμούς που γίνονται στα πλαίσια των διευθυντικών ταμείων, κάτι το οποίο εμάς σήμερα δεν μας φαίνεται και πολύ φυσιολογικό. Και έχω και παράδειγμα. Ξέρετε τι μάχη δίνουμε για την Ολλανδική καλωδιακή εταιρεία, την Τράκα. Η, η γαλλική Nexons παρετήθηκε από την αγορά και σήμερα έχει έρθει μια κινέζικη εταιρεία η οποία ε, προσπαθεί, χρησιμοποιώντας ε, την ευρωπαϊκή τεχνολογία για τις οπτικές ίνες, να πάρει το διαγωνισμό αυτό. Με τον κύριο Ταγιάννη, λοιπόν, εσείς ε, πώς συνεργάζεστε. Εκείνος προτείνει να δημιουργηθεί μια αρχή που θα εξετάζει τις ξένες επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς στην Ευρώπη. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να έχω την άποψή σας για αυτό το θέμα. Δεν θα αναφερθώ στη χρηματοδότηση. Εσείς μιλήσατε για τη χρηματοδότηση και πολύ καλά, είναι σημαντικό. Ε, τα κεφάλαια κινδύνου ή το ταμείο, το σχετικό, όλα αυτά είναι πολύ σωστά και σας στηρίζουμε κυρία Επίτροπε. Όμως, τι συγκεκριμένες προτάσεις κάνετε εσείς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια της πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σοντή τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι συγητής για την αξιολόγηση του ευδόμου προγράμματος ε, πλαισίου. Το πρόγραμμα αυτό ε, το διαπραγματευτήκαμε πολιτικά το 2006 και αποτελεί μέρος αυτού που ονομάσαμε τότε αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Υπάρχουν τρία νέα στοιχεία σε αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο. Πρώτον, ότι η στρατηγική αυτή απέτυχε. Δεύτερον, δεύτερο νέο στοιχείο, Έχουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, με νέα όργανα, με μια νέα κομισιόν και το τρίτο νέο στοιχείο είναι η κρίση, η οικονομική κρίση. Το πρόγραμμα αυτό το διαπραγματευτήκαμε στην αρχή της κρίσης. Σήμερα το 2011 είμαστε στα μέσα της κρίσης και έχουμε και το 2012 και το 2013 μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα. Ρωτώ λοιπόν μήπως πρέπει να τροποποιήσουμε κάτι. Επίσης κύριε Επίτροπε θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσέγγισή σας λέτε ότι δίνετε σημασία στη γνώμη του Κοινοβουλίου. Εμάς αυτό πραγματικά μας αγγίζει, το θεωρούμε σημαντικό, γιατί μεταξύ μας υπάρχει πολιτική συνένεση, μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων, ώστε μαζί να φροντίσουμε τα έτη αυτά, 2011, 2012 και 2013, να αποτελέσουν χρήσιμα έτη για την τεχνολογία, για την επιστήμη, για την καινοτομία. Όλοι θεωρούν ότι αυτά αποτελούν στοιχείο ανταγωνιστικότητας από το οποίο μπορεί να υποφεληθεί η Ευρώπη. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτό που με θλίβει είναι το ότι τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν και εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορέσαμε να έχουμε μια συνολική αξιολόγηση, κράτη-μέλη δηλαδή και Ευρωπαϊκή Ένωση, τη κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την έρευνα. Το είπε στον πρόεδρο, βέβαια δεν φταίει. Οπότε το ζήτημα είναι μήπως πρέπει να εξευρωπαίσουμε ακόμα περισσότερο την έρευνα και τότε δεν χρειαζόμαστε μια σφαιρική αξιολόγηση. Άλλη ερώτηση. Μήπως ήρθε η στιγμή για κάποια μεγάλα θέματα που εντοπίστηκαν από τους αξιολογητές να εποφεληθούν από υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παγκόσμια αριστείες δηλαδή, για κάποια θέματα που έχουν εντοπιστεί, όπως είναι οι κλιματικέ αλλαγέ, η υγεία, η γύναση του πληθυσμού, η ενέργεια, η πυρηνική ασφάλεια, η βιομηχανία. Τέλος, απλοποίηση. Ήσασταν ε, μέλος στο ελεκτικό συνέδριο, κύριε Επίτροπε, οπότε βασιζόμαστε σε εσά. Οι προτάσεις σας προς το παρόν δεν φτάνουν. Θα δημιουργήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ομάδες εργασίας, η κυρία Καβό για παράδειγμα έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, ώστε στο δημοσιονομικό κανονισμό να σας προτείνουμε τροπολογίες για να βγούμε από αυτό το πρόβλημα που είναι η διοικητική περιπλοκότητα και να υπάρξει απλοποίηση, κάτι το οποίο όλοι επιθυμούν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Λάμπερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, που ήρθατε. Ξέρουμε ποιος είναι ο ενθουσιασμός σας για να πετύχει η πολιτική μας στην Ευρώπη. Δύο ερωτήσεις, μία από τους πράσινους, το περιμένετε, και μία άλλη. Λοιπόν, αυτή που περιμένετε από μας είναι οι ανησυχίες που εκφράζουμε όλοι εμείς για τα ποσά τα οποία πηγαίνουν στην Ίτερ για επιπλέον χρηματοδότηση. 750 εκατομμύρια επιπλέον πάνε στο πρόγραμμα Ίτερ για τα έτη 2012 και 2013 χωρίς να μιλάμε για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα πλαίσιο και στο πώς θα προχωρήσει. 700 εκατομμύρια δεν είναι πολλά για επιπλέον χρήματα και για κάτι το οποίο είτε μπορεί είτε μπορεί να μην ε, μας επιτρέψει να έχουμε αποτελέσματα σε 50 χρόνια. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε και δεν τα ρωτάω αυτά μετά από όσα έγιναν στην Ιαπωνία, αλλά διαχειριστικά, καθαρά, είναι μια σωστή απόφαση για να δαπανίσουμε τα χρήματα αυτά. Τώρα μια λιγότερο αναμενόμενη ίσως ερώτηση από μένα. Ας κοιτάξουμε λίγο μπροστά. Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι να έχουμε αριστεία και στο μέλλον, αλλά από την άλλη μεριά να υπάρξει περισσότερη συνοχή στην συμμετοχή και να φροντίσουμε ολόκληρη η Ευρώπη να είναι οικονομία της γνώσης, όχι μόνο μερική, ένα μέρος της. Οι πρώτες χώρες θεωρούν ότι έχουν μείνει λίγο απ' έξω. Δηλαδή, τι εννοώ, με, τα, με την περιφερειακή πολιτική 50 εκατομμύρια, όσα περίπου για το πρόγραμμα πλαίσιο, θα μπορούσαν να δαπανηθούν για θέματα που έχουν κάνουν με έρευνα και ανάπτυξη. Κάποιες χώρες έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν και να προλάβουν τους υπόλοιπους στο επίπεδο αριστείας. Ρωτάω λοιπόν πώς αποτελεσματικά δαπανώνται τα χρήματα αυτά και δεύτερον, αν κοιτάξουμε καλύτερα το πρόγραμμα πλαίσιο όπως και αν ε, ονομαστεί τελικά, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνέργειες που υπάρχουν ε, με τα χρήματα που πάνε από το Περιφερειακό Ταμείο ε, σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα πλαίσιο. Ευχαριστούμε. 11 έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε προτείνω να κλείσουμε εδώ τον κατάλογο των ομιλητών και συγχρόνως να αρκεστείτε σε δύο λεπτά ο καθένας, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Ο κύριος Φανίστερο τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Ήδη τα πάνε και οι συνάδελφοι πόσο σημαντικό είναι να δούμε σε διεθνές επίπεδο την πολιτική μας και την στρατηγική μας και τα συμφέροντά μας. Φυσικά και χρειάζεται συνεργασία για την αριστεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εννοείται. Όμως υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται από την κινέζικη κυβέρνηση για παράδειγμα για την γνώση από την άλλη μεριά δικές μας επιχειρήσεις ε, μετακινούνται, μεταφέρονται αλλού. Δεν θα έπρεπε να το δούμε αυτό. Δεύτερον, για τα ταμεία, για τα χρήματα από το Περιφερειακό Ταμείο προς την Ανατολική Ευρώπη, που είπε και ο συνάδελφος. Εγώ βλέπω να υπάρχει μια θετική εξέλιξη, γιατί κοιτάξτε τι γίνεται στην Πολωνία, στην Τσεχία. Όντως, πρέπει η αριστεία αυτή να καλύψει και αυτούς με επενδύσεις βέβαια συγχρόνως στις επενδύσεις παντού. Έχω και μία παρατήρηση για το Facility Fund. Όταν αποφασίσαμε για τα δισεκατομμύρια αυτά για το πρόγραμμα πλαίσιο δεν ήταν και για την έρευνα και τις υποδομές. Μήπως κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω. Οπότε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι η μεγάλη επένδυση πώς θα γίνει. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερο output. Κατάλαβα ότι υπάρχει το Συμβούλιο το οποίο βέβαια αποφασίζει, αλλά θα προσαρμοστούν τα κριτήρια ή θα συνεχίσουμε με τα ίδια κριτήρια παρόλο που ξέρουμε ότι δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Και τέλος μια ερώτηση για σας για την καινοτομία και το έγγραφο που υπάρχει. Λέει ότι μία φορά το χρόνο θα οργανώνεται μία συνέλευση για αυτό το θέμα. Το 2011 ήδη μπορεί να υπάρξει μια τέτοια τροπολογία, ε, συγγνώμη, πρωτοβουλία η οποία έρχεται και από το Κοινοβούλιο. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν. Ένσου. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω την Επίτροπο σήμερα το πρωί και να της ευχηθώ κάθε επιτυχία μετά από όσα έγιναν στις 7 Μαρτίου. Να πω την άποψή μου για το μέλλον της έρευνας και της κοινοτομίας. Νομίζω ότι στο πρόγραμμα πλαίσιο έχουμε τη δυνατότητα για περαιτέρω ε, δραστηριότητα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση των νέων προϊόντων στην αγορά θα είναι ταχύτερη. Θα δημιουργηθεί περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συναρμοστεί με την βιομηχανική μας πολιτική. Μιλώντας τώρα για την ε, συνοχή και τη σχετική αναθεώρηση. Σε πολλέ συζητήσει έχω υπογραμμίσει ότι κάποια από τα νέα κράτη-μέλη δεν έχουν τις απαραίτητε ερευνητικέ υποδομέ. Εσεί εσείς είπατε ότι ειδικά κονδύλια θα μπορούσαν να αφοσιωθούν ε, σε αυτό το στόχο. Στην επιτροπή μα χθε συζητήσαμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματο πλαισίου για την έρευνα και με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, του κυρίου Ρόλφ Άνεμπεργκ. Όταν το ρώτησα το ίδιο πράγμα, μου είπε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διευθυντικά ταμεία για αυτό το στόχο. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα σωστός τρόπος να εξεύρουμε νέα χρηματοδότηση, επιπλέον χρηματοδότηση για τα νέα κρατημέλη. Ξέρω ότι υπάρχει σοβαρό ανταγωνισμό μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και των υπόλοιπων ε, χωρών, όπω ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική Λογουχάρη και τα κράτη-μέλη διμερό. Και όχι μεταξύ των κρατών μελών αυτών καθεαυτών. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Επίτροπο για τη σημερινή της παρουσία. Με μεγάλη προσοχή άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι θα εστιαστώ στα βαθιά πολιτικά ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Σοντή, γιατί νομίζω ότι η συζήτηση σχετικά με το πού πάει η Ευρώπη σε σχέση με την έρευνα και την καινοτομία, με τη βασική υπόθεση εργασίας, ότι αυτό είναι ο δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτοχρόνως η Ευρώπη μαστίζεται από μια μεγάλη οικονομική κρίση, και ταυτοχρόνως το παγκόσμιο σκηνικό και η ισορροπία της ανάπτυξης μεταφέρεται από τη Δύση προς τον Ειρηνικό και την Ασία, θα ήθελα να θέσω δύο-τρία ερωτήματα συναφή προς αυτά που έθεσε ο κύριος Οντή. Καταρχήν πρέπει να δηλώσω ότι ενοχλούμε από τον αυτιστικό τρόπο που η Ευρώπη εξετάζει το μέλλον της. Θα ήθελα να μας είχαν παρουσιαστεί στοιχεία που δείχνουν και είμαι βέβαιος ότι τα έχετε εσείς στη διάθεσή σας κυρία την σχετική θέση της Ευρώπης σε σχέση με τον παγκόσμιο γίγναστο. Δεύτερον, δεν μπορούμε να προσπερνάμε την αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας και να οραματιζόμαστε το όραμα του 2020 χωρίς να έχουμε καταλήξει συμπέρασμα τι έγινε και γιατί αποτύχαμε στη στρατηγική της Λισαβόνας. Έχουμε πάρει πάρα πολλές αποφάσεις δεσμευτικού τύπου για ό,τι πράγματα θέλετε, για τις ανανεώσιμες, για την ενέργεια και ούτω καθεξής. Θα μπορούσαμε άραγε να πάρουμε μια δεσμευτική απόφαση έτσι ώστε η κρατική επιχορήγηση υποχρεωτικά να γίνει 1% μέχρι το 2015. Το ζήτημα της συνοχής, το ζήτημα των διαρθρωτικών ταμείων είναι και πάλι βαθιά πολιτικό ή πιστεύουμε στην αριστεία ή πιστεύουμε στη συνοχή. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ιδρύσει ένα μηχανισμό στήριξης όπως ακριβώς στην οικονομία για να βοηθήσει τα αδύναμα κράτη που δεν τα καταφέρνουν στην έρευνα με δική της παρέμβαση στη διαχείριση των διευθυντικών ταμείων για την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλοι κύριε Δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να δούμε λιγάκι ένα κεντρικό σημείο στις εργασίες μας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η αναθεώρηση του προηγούμενου προγράμματος πλησίου έχει δύο συνέπειες. Η μία είναι μεσοπρόθεσμη, δηλαδή τι πτυχές της αναθεώρησης αυτής τι είναι σημαντικέ προκειμένου να τι λάβουμε υπόψη μας και να τις εφαρμόσουμε όταν σχεδιάσουμε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και κάτι άλλο είναι βραχυπρόθεσμο και αυτό είναι στην πράξη άμεσα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε στο χρόνο που μένει για το πρόγραμμα αυτό πλαίσιο που ολοκληρώνεται το 2013 τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη συνέχεια αυτή. Πολλέ φορές βλέπετε συζητάμε για θέματα τα οποία δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογή. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα τα οποία δεν εγκρίνονται για το 2011 για το 2012 για παράδειγμα. Συνεπώς, τι δυνατότητε υπάρχουν σε πολλές από τις πτυχές ε, που συζητάμε να ξέρουμε ότι άμεσα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Από την άλλη, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ό,τι μένει από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Τώρα και στην έκθεση των ειδικών. Αναφέρονται διάφορα πράγματα από τα οποία εσείς ποια πιστεύετε ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό που μένει από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πώς μπορεί να υποφεληθεί το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο από την αξιολόγηση που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι πιστεύω ζωτική σημασία γιατί είναι στην πράξη πώς θα χρησιμοποιήσουμε την αξιολόγηση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Καρβάλιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την παρουσία της σήμερα εδώ. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά την απλούστευση. Καλωσορίζουμε τα μέτρα που ήδη έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω όμως ότι απομένουν μέτρα και στην ανακοίνωση τη Επιτροπή αναφέρονται και στη δική μου την έκθεση που θα μπορούσαν να εκτελεστούν χωρί να, να, να αλλάξει ο δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό νομίζω αναφέρεται και στην, ενδιάμεση, στην έκθεση ενδιάμεσης αναθεώρησης για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Την έκθεση αυτή άλλωστε και σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού την εξετάζει η Κοκομπού, η Επιτροπή των Προπολογισμών. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε το ανεκτό επίπεδο σφάλματος ή κινδύνου. Θα πρέπει να αναζητήσουμε έναν τελείως καινούριο τρόπο για να αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, ώστε να επιτρέψουμε περαιτέρω έρευνα και σε μεγάλα και σε μεσαία προγράμματα. Ήθελα λοιπόν τη δική σας άποψη σχετικά. Ένα δεύτερο σχόλιο. Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία της αναθεώρησης του 7ου προγράμματος πλαισίου όπως είπε και ο συνάδελφος Οντή, ώστε να αλλάξουμε όσα χρήζουν αλλαγή. Εδώ κάποια στοιχεία στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν πολύ θετικά. Καλό είναι να τα διατηρήσουμε. Όμως και στις θεματικές προτεραιότητες θα πρέπει να προσαρμόσουμε ό,τι χρήζει προσαρμογής. Λόγω χάρη η ενέργεια δεν ήταν για την ώρα μεγάλη προτεραιότητα όταν σχεδιάστηκε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό και στην βιομηχανία. Και επίση και στη διάρθρωση και του μηχανισμού. Υπάρχουν στοιχεία που καλό θα ήταν να αλλάξουν. Θα πρέπει λόγω χάρη τα GTI να είναι πιο ανοιχτά σε πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να επανασχεδιάσουμε τα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλήσατε για την συμμετοχή των γυναικών επίσης. Διερωτώ με, δεν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές επιστήμονες και επιστημόνισες. Έχουμε πολλές τέτοιες στη χώρα μου, ε, την Πορτογαλία, οι οποίες βρίσκονται άνεργες. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να τους δώσουμε κίνητρα, ώστε να μπορούν να είναι ενεργοί συμμετέχοντες σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Ευχαριστούμε κυρία Κόμη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για τα όλα αυτά που μας είπε γιατί ήταν πάρα πολύ χρήσιμα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πράγματι πρέπει να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία γιατί είναι ένα θέμα κλειδί. Παράλληλα όμως θεωρώ ότι οι νέοι ερευνητές και οι ερευνήτριες ε, κυρίως ε, είναι ένα ε, θέμα που επίσης έχει μεγάλη σημασία και θέλω να προτείνω ίσως ε, οι νέες ερευνήτριες ε, οι οποίες στη δική μου την περίπτωση είναι οι, οι λιγότερο εκπροσωπούμενοι κατηγορίες αυτές θα μπορούσαν να προωθηθούν περισσότερο. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο διότι η Ιταλία, η χώρα μου, είναι μια χώρα η οποία δεν επωφελείται επαρκώς από τη χρηματοδότηση και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Ευρώπη αυτό είναι περισσότερο ένα θέμα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Ε, τώρα, κάτι άλλο. Ε, θέλω ε, να σας ρωτήσω εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα ισορροπήσετε την καινοτομία με την εφαρμοσμένη έρευνα γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα κλειδί που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίπλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να θίξω δύο θέματα. Καταρχήν και σας ε, ευχαριστώ πολύ και σας ε, κύριε Επίτροπε και που ήρθατε και για όλα αυτά που μας είπατε. Έχοντας κατά νου την καταστροφή στην Ιαπωνία, ρωτώ λοιπόν... Ε, προβλέπετε ε, να επεκτείνετε, την, ε, να ασχολείται περισσότερο με την τεχνολογία που έχει σχέση με την ενεργική ασφάλεια, τα θέματα της ε, μπαταρίας, πολλά θέματα που άπτονται αυτού του τομέα. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω κυρία Επίτροπε, έχει σχέση με τις επιστήμες πνευματικής ιδιοκτησίας και κατεύθυνσης, γιατί υπάρχουν φήμες ότι αυτές οι επιστήμες δεν θα τύχουν στο μέλλον της ίδιας υποστήριξης. Εγώ αυτό το θεωρώ λάθος και θα ήθελα να ακούσω από εσά έτσι μια πρώτη αντίδραση, κατά πόσον ε, συμφωνείτε κι εσείς με τους άλλους ή με συντάσσεστε περισσότερο με τη δική μου άποψη. Πρόεδρος, το πρόβλημά μου είναι ότι έχουν ζήσει το λόγο άλλοι δύο-τρεις συνάδελφοι. Ε, οι οποίοι ήρθαν λίγο αργότερα. Εμεί όμω είχαμε αποφασίσει να κλείσουμε τον κατάλογο των ερωτώντων και αυτό τώρα για μένα είναι πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει αποφασίζω τώρα θα παραμείνω στον κατάλογο που είχα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κυρία Επίτροπε. Έχω ορισμένε ερωτήσει για τη σχέση μεταξύ τη Ένωση για την Κοινοτομία και του προγράμματο πλαισίου. Μπορείτε να μα πείτε κατά ποιον τρόπο αυτή η Ένωση μπορεί ή όχι να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για το πώς θα εξελιχθεί το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Και εδώ μιλήσατε για προκλήσεις, βασικές προκλήσεις. Αυτές οι προκλήσεις θα μπορούσε να είναι επίσης ένα ζωτικό στοιχείο για το πρόγραμμα πλαίσιο. Εάν μπορούσαμε να εντοπίσουμε δύο τέτοιες βασικές ε, προκλήσεις ή τρεις. Πώς θα τις αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτές τις προκλήσεις θα τις συσχετίσετε με την έρευνα ή θα τις χωρίσετε σε ομάδες. Επίσης για τις εταιρικέ σχέσεις για την καινοτομία. Πώς θα ευθυγραμμιστούν με το πρόγραμμα πλαίσιο. Όλα τα στοιχεία του προγράμματος πλαισίου πρόκειται να εφαρμοστούν ε, βάσει σχέσεων εταιρικής, βάσει εταιρικών μάλλον σχέσεων. Εμένα με ανησυχούν κάπως αυτές οι εταιρικέ σχέσεις. Παντού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να υπάρχουν τέτοιες σχέσεις εταιρικέ καινοτομία. Είναι σαν να βρήκαν όλοι ένα καινούργιο εργαλείο ξαφνικά και το χρησιμοποιούν διαρκώς. Αλλά εμείς ως κοινοβούλιο δεν μπορούμε να το καλύψουμε αυτό ακόμη. Δεν έχουμε δικαίωμα άποψης εδώ, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τι ε, εννοούν λοιπόν αυτές οι εταιρικές σχέσεις. Και επίσης πού θα δοθεί έμφαση στο πρόγραμμα πλαίσιο. Εδώ σε τι θα δώσουμε προτεραιότητα και σε τι θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει αρνητική προτεραιότητα. πως θα το κάνετε λοιπόν εσείς αυτό, θα δείτε μόνο τις προτεραιότητες θα δείτε και τις αρνητικές προτεραιότητες Οι προκλήσει, εφόσον αυτές θα οδηγήσουν ε, την πορεία που θα ακολουθήσουμε, τι θα αφήσετε κατά μέρος και για τους πολίτες μας που είναι πολύ σημαντική για αυτούς η καινοτομία. Ε, πώς θα καλυφθεί η ανάγκη αυτή στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και έπειτα για τη χρηματοδότηση. Θα μετατοπίσετε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης στο κοινό κεφάλαιο κινδύνου. Ο κύριος Γκίρεκ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εδώ δεν θέλω να διαφρονικήσω μαζί σας για την έννοια της αριστείας. Ο καθένας μπορεί να είναι άριστος, όμως είναι μια έννοια τελείως υποκειμενική, η οποία για ορισμένες επιστημονικές κοινότητες υπονοεί ε, κάποιες αδιαφανείς ε, αρχές. Δεν ξέρουμε πώς γίνεται η κατηγοριοποίηση, ούτε πώς γίνεται η επιλογή των σημαντικότερων προβλημάτων ε, που εξετάζονται. Εδώ υπάρχει θέμα με την προβολή. Τα εργαλεία που επιλέγονται, τις μεθόδους, δεν είναι πάντοτε τα καλύτερα. Πιστεύετε ότι αυτή η προσέγγιση είναι σωστή. Πιστεύετε ότι η επιστημονική δυνατότητα, το επιστημονικό δυναμικό της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αξιοποιείται παρκώς. Θα πρέπει νομίζω αυτή την αρχή να την αντικαταστήσουμε με τις πραγματικές δυνατότητες που διαθέτουμε, όπως λόγου χάρη είχε γίνει με συγκεκριμένα προγράμματα στο παρελθόν. Ευχαριστούμε κυρία Μαντουρέλου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο που ήρθε για να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί όσον αφορά το μέλλον της επιστημονικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντα υπόψη βέβαια και την καινοτομία. Πολύ σύντομα θα ήθελα να σας μεταφέρω μία ανησυχία μου. Συμφωνώ μαζί σας για το ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρη η στόχη και το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στους πολίτες μας. Και ένα από τα σαφή μηνύματα που πρέπει να περάσουμε είναι εκείνο της ισορροπίας. Και δεν ξέρω αν το πετυχαίνουμε. ισορροπία εννοώ βασική έρευνα, θεμελιώδης και καινοτομία. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ανισορροπία ήδη. Έπειτα συνέχεια, όσον αφορά τη συνέχεια που δίνουμε σε ό,τι πήγε καλά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και τα νέα μέσα που είναι αναγκαία για να πετύχουμε καινούριου στόχους. Αν δεν υπάρχει μια ελάχιστη συνέχεια, δημιουργείται αβεβαιότητα. Χρειάζεται επίσης ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη που δίνουμε στις ερευνητικές ομάδες που κάνουν ένα πάρα πολύ καλό έργο, αλλά συγχρόνως και στήριξη στους νέους ερευνητές. Και αυτό βοηθάει να δώσουμε σιγουριά στους πολίτες μας και να αποφύγουμε ε, φόβους που λένε ότι προσπαθώντας να βελτιώσουμε κάποια πράγματα μειώνουμε το συνολικό προπολογισμό. Έπειτα χρειάζεται και ισορροπία στην αύξηση των ε, ερευνητών, δηλαδή στην αναλογία που υπάρχει ανακάτοικο, έτσι ώστε να πετύχουμε μια καλή αναλογία όπως έχουν οι χώρες που μας ανταγωνίζονται. Αν πετυχαίναμε όλες αυτές τις ισορροπίες θα καθησυχάζαμε και τους ερευνητές αλλά και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στα θέματα της έρευνας και της τεχνολογίας και της καινοτομίας για το μέλλον της έρευνας και για το μέλλον της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Σίγουρα το γνωρίζει και η Επίτροπος. Υπάρχουν διάφορες διαδόσεις που κυκλοφορούν. Αυτή ακριβώ είναι η ανησυχία μου. Και ήθελα να σας τη μετεφέρω ώστε να φροντίσετε να κάνετε κάτι για να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδόσεις και τέτοιου είδους ανησυχίες μεταξύ των πολιτών μας. Η κυρία Τόγια. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ ε, θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Επίτροπε για την σαφήνεια της παρουσίας σας και το πάθος που δείχνετε για όλα αυτά τα θέματα και για τις αρμοδιότητες σας γενικότερα. Εδώ ήθελα να περάσω σε ένα θέμα ουσίας, αφορά τους πόρους. Είναι πλέον σαφές για όλους ότι υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ των στόχων της, ε, των προτεραιοτήτων της στατικής το 2020 και των πόρων των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Μιλάμε εδώ για κονδύλια τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε μέσα από τις προσπάθειές μας και που κινδυνεύουν να φέρουν έλλειψη ισορροπίας στο όλο μας σύστημα. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, μιλήσαμε εδώ για την πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ταγιάννη, υπάρχουν πολλές επενδύσεις που έρχονται από άλλες χώρες, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος, χωρίς διαφάνεια. Έτσι λοιπόν Νομίζω το θέμα αυτό πρέπει να το εξετάσουμε και από την πλευρά των επιτρόπων που κοιτάζουν την ουσία του θέματος. Με ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα η εξέταση του θέματος από την Επιτροπή Κρίς, ε, η οποία, ε, όπως είπε και ο ένα συνάδελφο, ε, μα αναγκάζει όλοι εξέταση του θέματο των κονδυλίων να δούμε μια σοβαρή ανάγκη. Πόσα είμαστε πρόθυμοι να εκταμιεύσουμε, να δραστηριοποιήσουμε για να φτάσουμε του στόχου μα. Για τον προπολογισμό λοιπόν μέχρι το 2020 Ποιο είναι ο στόχο να διατηρήσουμε του πόρου σταθερού, όπω ε, όπως προβλέπονται στον προπολογισμό. Όμω για το μέλλον πρέπει να κάνουμε κάποιο θετικό βήμα. Νομίζω λοιπόν Όπω λένε όλοι, ότι εδώ πρέπει να αναζητήσουμε εργαλεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλή. Δεν μπορούμε εδώ με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό να περιμένουμε ότι θα ενισχυθούμε περαιτέρω από τα εθνικά κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν τα διάφορα οικονομικά εργαλεία που διαθέτουμε στο συγκεκριμένο τομέα να τα δραστηριοποιήσουμε για να κατανείμουμε τον κίνδυνο, να αναζητήσουμε επενδύσει, περαιτέρω κονδύλια. Μιλήσαμε και για το εργαλείο διευκόλυνση για την κατανομή του κινδύνου, το σχολιάσετε, αλλά θα πρέπει ενδεχομένω να αναζητήσουμε και νέα εργαλεία, τα οποία ακριβώ να μπορούν να λειτουργήσουν ω πολλαπλασιαστέ των κονδυλίων. Αυτό λοιπόν είναι καθοριστική σημασία. Πρέπει να ενώσουμε τι προσπάθειέ μα για να κάνουμε σωστή δαπάνη κάθε ευρώ του προπολογισμού, για να χρησιμοποιούμε την προστεθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Συμβολή, για να συσχετίζουμε με τα ταμεία συνοχή, για να βρίσκουμε όλε τι δυνατότητε διασυνδέσει, για να κάνουμε ένα κοινό προγραμματισμό. Αυτέ οι προσπάθειε όμω θα είναι επαρκεί εάν δεν δούμε πόσο η μεγάλη εμβέλεια έχει αυτή η πρόκληση που αφορά την καινοτομία και την έρευνα γενικότερα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ähm, ich will mal ein Stück weg von der Sachdiskussion. Εγώ θα ήθελα λιγάκι να, πω, να φύγω λιγάκι το θέμα και να πω το εξή ότι αν τελικά ε, δώσουμε 20% περισσότερα για το ε, ερευνητικό πρόγραμμα 8, τότε <clears throat> κατ' ουσίαν μόνο μέχρι το καλοκαίρι έχουμε χρόνο για να συνάψουμε το συμβιβασμό εκείνο που θα μας επιτρέψει ε, να ε, επιτύχουμε το στόχο μας. Πρόκειται για συμβιβασμό ανάμεσα στα παλιά και στα νέα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες, αλλά να πω το εξή. Αν δεν καταλήξουμε σύντομα σε συμβιβασμό, τότε θα συμβεί αυτό που διαφαίνεται. Δηλαδή, θα έχουμε μια δύσκολη ε, δημοσιονομική και κατάσταση και κατάσταση προπολογισμού τα νέα κρατημέλη φοβούνται την αριστεία και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον μάλλον τα παλιά, τα παλιά θα φοβούνται την αριστεία, αλλά και τα νέα ε, θα ε, θέσουν ένα αμφιβόλο θέματα όπως είναι το πρόγραμμα Γκαλιλαίο και άλλα. Πρέπει λοιπόν αρκετά νωρίς ε, να βρούμε ένα συμβιβασμό. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό έγκαιρα, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ότι δεν θα υπάρξει σημαντική αύξηση των κονδυλίων χρηματοδότησης. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω ε, το συντομότερο δυνατόν και μάλιστα ίσως και στην πράσινη βίβλο ε, να καταλήξουμε σε μια έτσι γενική διαπίστωση ε, και όταν θα μιλάμε για το πολιετές πλαίσιο ε, τότε θα συζητηθεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο μέχρι το τέλος του έτους. Και μέχρι τότε, αν δεν έχουμε ένα αίτημα που θα είναι τουλάχιστον αύξηση κατά 20 25% των κονδυλίων. Δεύτερον, συμβασμό σε αυτό το κέριο θέμα, αν δεν τα κάνουμε αυτά, τότε για διάφορους λόγους τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο θα επικρατήσει διχασμός και αποτέλεσμα αυτού δεν θα υπάρξουν επιπρόσθετα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν εγώ τάσομαι αναμφίβολα ε, υπέρ του ε, πολιτικού μηνύματος ε, να δρομολογήσουμε το συμβασμό γιατί αλλιώ θα χάσουμε τη μάχη. Στο πρόγραμμα των υπαριθμών 7 συζητάγαμε μέχρι τέλους αυτά τα θέματα και αυτό ήταν μια μεγάλη αδυναμία μας γιατί αν δεν βρούμε το συμβασμό έγκαιρα στο τέλος εκεί τι έγινε, υπήρχε ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια και με μεγάλο κόπο τα ανακτήσαμε ε, και μπορέσαμε έτσι να έχουμε μια συμβολική αύξηση κονδυλίων. Τέλος όμως με αυτό. Τώρα πια θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο έξυπνα, να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη ποια είναι η ακριβής αύξηση των κονδυλίων που διεκδικούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η τελευταία ερώτηση από τον κατάλογο των ερωτώντων. Έχουμε άλλα 10 λεπτά και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να προσπαθήσει να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα που δεν είναι εύκολο στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει διαθεσή τη, αλλά μπορεί να απαντήσει τα σημαντικότερα. Παρακαλώ, το Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετά για να απαντήσω σε όλα αυτά τα ερωτήματα, αλλά θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω. Πρώτα απ' όλα, αυτό το θέμα που διαρκώ επανέρχεται για την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματο πλαισίου και το ποιε είναι οι διαφορέ μεταξύ των χωρών που τα πάνε πολύ καλά και των χωρών που δεν έχουν την ίδια προοπτική Νομίζω ότι ευθύ εξ αρχή πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αυτή εξ αρχή από την αρχή λειτουργία δηλαδή του 7ου προγράμματο πλαισίου έχουμε κάνει σοβαρέ προσπάθειε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Και αυτό σημαίνει ότι ενεργώ προσπαθούμε να προσλάβουμε ανεξάρτητου ελεγκτέ από ολόκληρη την Ευρώπη, διατηρώντα την αρχή τη αριστεία. Διατηρήσαμε τα εθνικά σημεία επαφή. και των νέων και των παλιών κρατών μελών και μας ανησυχεί ότι υπάρχει, υπάρχουν διαρκώς αρνητικά αποτελέσματα κάποιων που δεν φτάνουν τους υπόλοιπους παρά μόνο πολύ δύσκολα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορεί να οδηγούν και στην στα αρνητικά αποτελέσματα, στι χαμηλέ επιδόσει, και αυτό το παρακολουθούμε. Βρισκόμαστε στη φάση τη ε, παρακολούθησης του γιατί συμβαίνει αυτό. Ακούμε μέσω τη πράσινη βίβλου και προσπαθούμε να ακούσουμε και του ειδικού για να μάθουμε από τι απόψει του. Βεβαίω, κάποια σημεία εδώ και από τα διαφορετικά ταμεία είναι πολύ σημαντικά γιατί χρειαζόμαστε τι εξαιρετικέ ε, υποδομέ έρευνα των χωρών που του λείπουν. Οι βουλευτέ και οι υπουργοί από τι χώρε αυτέ, διαρκώ μου λένε ότι έχουν του καλύτερου ερευνητέ, του καλύτερου επιστήμονε φεύγουν από τι χώρε αυτέ, πάνε να δουλέψουν αλλού ε, και όχι μόνο σε ευρωπαϊκά κράτη, κάποιοι πάνε ανατολικά και κάποιοι δυτικά. Και αν έχουμε τι εξαιρετικέ υποδομέ που θέλουμε για την έρευνα, αυτό μπορεί να μην συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά τεχνολογία. Βεβαίω, εδώ μα ενδιαφέρει μια αμφίδρομη σχέση που θέλουμε να δημιουργηθεί με τι ε, αναδυόμενε οικονομίε και χώρε. Έχουμε υψηλό επίπεδο διαλόγου ε, με την Κίνα, όπως ξέρετε, χάρη στην σχετική ομάδα, την αρμόδια ομάδα. Ξεκίνησε συζήτηση από πέρσι και στο Πεκίνο φέτος είχαμε συνάντηση. Εγώ ίδια θα επισκεφθώ την Κίνα αργότερα φέτος και αυτό το θέμα πρόκειται να το θέσω. Θα το θέσω γιατί είναι πρώτης προτεραιότητας για όλους στην, στο δυτικό κόσμο, αλλά ιδίω για εμάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση. Συνεχώς Αναφέρω την εξαιρετική έκθεση της ε, βουλευτού Μαρία Καρβάλιο, γιατί πραγματικά αποτελεί το θεμέλιο για όλα τα μέτρα απλούστευσης, τα οποία πρέπει να προβλέψουμε. Το έχω πει επανειλημμένως όλα τα μέτρα απλούστευσης που μπορούμε να προβλέψουμε αυτόβουλο από την πλευρά της Επιτροπής έχουν ήδη προβλεφθεί. Είναι στα δικά σας χέρια το όλο θέμα και στα χέρια του Συμβουλίου για να προχωρήσει το θέμα όπως είπε η κυρία Καρβάλιο. Χρειάζονται και άλλα μέτρα απλούστευσης ε, μέσα από τις αναθεωρήσεις του προπολογισμού και του ε, TRE. Διότι όταν ψήφισε η Ολομέλεια την έκθεση Καρβάλιου, ε, αυτό ήταν μέρος της όλης προσπάθειας απλούστευσης. Ε, Εμεί καταλαβαίνουμε λοιπόν με την ψηφοφορία τη Ολομέλεια ότι το κοινοβούλιο μα στηρίζει, μα λέει να πάμε μπροστά. Αυτό και θα κάνουμε λοιπόν, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προ αυτή την κατεύθυνση. Προφανώ τέθηκε το θέμα Twitter. Εδώ το έχω πει και αυτό επανειλημμένο και το γνωρίζει ο κύριο Λάμπερτ πολύ καλά. Εδώ αυτό το θέμα για μένα αποτελεί ένα δύσκολο θέμα μετά την ψηφοφορία του περσινού προπολογισμού, όπου δύο τρίτα τη χρηματοδότηση προέρχονταν από άλλου πόρου και ένα τρίτο μόνο από το πρόγραμμα πλαίσιο, είχαμε βρει μια προσωρινή λύση. Το είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Όμω είχε γίνει τεράστια, τεράστιο θέμα διαφιλονικία μεταξύ Γενική Διεύθυνση και δική μου τοποθέτηση για το να μην ξεπεράσουμε αυτό το ένα τρίτο. Ξαναήρθε η συζήτηση για τον προπολογισμό, όμω και είδατε ότι έχουμε πέσει θύματα τη παγίδα αυτή τη απόφαση τελικά για το ΙΤΕΡ. Κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί εδώ μια λύση. Νομίζω ότι είναι αποφασιστική σημασία να βρεθεί τέτοια λύση, διότι οι συνέπειε για τι χώρε που τώρα έρχονται και οι εταιρείε που τώρα υπογράφουν συμβάσει πρέπει να διευκολυνθούν. Το, το εργαλείο διευκόλυνση δεν επιλογού χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ευοδοθεί. Εδώ νομίζω η κυρία Νίμπλερ έθεσε ένα θέμα και σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία τις τελευταίες ημέρες. Αργότερα σήμερα θα συναντηθούμε με τον Επιτρόπο Έτιγκερ που έχει ε, αρμοδιότητες εδώ για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και θα συζητήσουμε. Δεν νομίζουμε ότι άμεσα υπάρχουν συνέπειε για του Ευρωπαίου. Τα επίπεδα ραδιενέργεια, ε, είναι στα φυσιολογικά επίπεδα για τα κράτη-μέλη τουλάχιστον. Μέτρα ε, είναι διαρκώ σε λειτουργία και τα διάφορα κράτη-μέλη με του σταθμού μέτρηση τη ραδιενέργεια στην επικράτειά του, τα παρακολουθούν. Επίση, η Επιτροπή χρησιμοποιεί το σύστημα Curie που είναι σύστημα μέτρηση και προειδοποίηση, και στην περίπτωση που η ραδιενέργεια ξεπερνά κάποια ανεκτά επίπεδα σε ένα κράτο μέλο, όλοι ειδοποιούνται αμέσω. Όμω, τα κράτη-μέλη έχουν και οι ίδιοι ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη και για τι άδειε που δίνουν στου διάφορου ε, παράγοντε, καθώ και τη συμμόρφωση αυτών με τι απαιτήσει ασφάλεια. Φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου θα έχουν πολλά να πούν γι' αυτό. Ο ρόλος ε, του Κοινοβουλίου στις ε, διάφορες ε, εταιρικέ σχέσει αναφέρθηκε ήδη. Εδώ έχουμε συμμετοχή των βουλευτών και εκπροσώπων του Κοινοβουλίου στι ομάδε που ασχολούνται με το θέμα τη γύρανση του πληθυσμού. Νομίζω ότι θα αποσταλεί πρόσκληση και στον πρόεδρο Μπούζεκ απευθεία για να φροντίσει την εκπροσώπηση και γενικότερα για τι EIP. Πρέπει να πω ότι είχαμε σοβαρότατη συζήτηση ευθύ εξ αρχή και εδώ και στο Συμβούλιο. Ιδίω σε ό,τι αφορά τη ίδια τη εταιρική σχέση. Αποφασίσαμε να έχουμε μια πιλωτική φάση σε πρώτη φάση. Το Συμβούλιο αρχικά παρακολούθησε το θέμα και τελικά μας έδωσε και το πράσινο φως για την πιλωτική φάση. Αυτή η πιλωτική φάση ω τέτοια θέλουμε να λειτουργήσει. Να δούμε ακριβώς τι θέλουμε να γίνει με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ε, ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις για την καινοτομία. Εφόσον δοκιμαστούν και πετύχουν θα προχωρήσουμε, Όπω και εσεί, κυρία Μέρκη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τόσοι πολλοί συνάδελφοι θέλουν τέτοιε εταιρικέ σχέσει καινοτομία. Όμω έχουμε αυστηρότατα και θα γίνουν ακόμη πιο αυστηρά τα κριτήριά μα σε σχέση με το τι σημαίνει ευρωπαϊκή σχέση, εταιρική σχέση καινοτομία. Ε, Βεβαίω μα περιορίζει το γεγονό ότι πρέπει να ξαναπάμε στο Συμβούλιο για έγκριση πριν ανακοινωθεί η έναρξη του επόμενου σταδίου. Είμαστε λοιπόν στη φάση της δοκιμής. Χρειάζεται τέτοιου είδους υλοποίηση για όλου αυτού του, την ομάδα πρωτοβουλειών. Νομίζω επίσης, πολύ σωστά, πολλοί βουλευτές ανέφεραν τις περιφέρειες. Ξέρετε ότι οργανώνουμε διάσκεψη των περιφερειών στι Βρυξέλλε τον Ιούλιο και το θέμα θα είναι πόσες περιφέρειες περιφερειέ μπορούν να αποφεληθούν από τα 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την διάσκεψη αυτή, διότι οι περιφέρειες και επειδή εγώ είχα την ευκαιρία να τι επισκεφθώ στα διάφορα κράτη-μέλη, μα είπαν δεν γνωρίζουμε αρκετά. Δεν ξέρουμε τι διατίθεται. Θέλουμε να συμμετέχουμε κι άλλο. Για το RSFF. Εδώ αναζητούμε ένα ευρωπαϊκή εμβέλεια εργαλείο, ακριβώς στα πλαίσια αυτού του εργαλείου της ε, διευκόλυνσης ε, για την ε, κατανομή του κινδύνου στην έρευνα. Προσπαθούμε εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να ζητούμε νέα δημοσιονομικά εργαλεία ώστε να καλύψουν κάποιε από τι μέρημνε που ανέφεραν και τα μέλη τη Επιτροπή σα. Βεβαίω, στην Επιτροπή αυτή περιλαμβάνεται και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που μας λένε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να βοηθήσουν για να ανακουφίσουν από το πολύ μεγάλο οικονομικό βάρος που θα συνεχίσει να ασκείται και στο μέλλον στον προπολογισμό. Ως προς το μελλοντικό λοιπόν προπολογισμό βρισκόμαστε απολύτως στα χέρια του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εδώ έχω συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένω τη στήριξη, τη συμπαράσταση των μελών τη δική σα τη Επιτροπή για τα όσα αφορούν την έρευνα και την κοινοτομία. Συγκεκριμένα, για την επαναδιοργάνωση της γενικής μας διεύθυνσης. Δεν θέλω κανείς να φύγει από εδώ με την εντύπωση ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες θα παραμεληθούν και ότι υπάρχουν ερευνητικά στοιχεία στα οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι σε άλλα. Μην φύγετε με αυτή την εντύπωση. Έχουμε συνέστηση και σκοπεύουμε να στηρίξουμε όλα τα στοιχεία. Βεβαίω το κοινό στρατηγικό πλαίσιο θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις γενικότερες προκλήσεις ε, της κοινωνίας των εταιριών. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις πρέπει κυρίως να επικεντρωθούμε στην βασική έρευνα. Λύσεις σε αυτές τις βασικές προκλήσεις δεν μπορούμε να βρούμε αν δεν έχουμε τις βέλτιστες, τις πλέον άριστες ε, ερευνητικές λύσεις. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για όλες τις ερωτήσεις και με συγχωρείτε που είχα τόσο λίγο χρόνο. Ελπίζω ότι θα, θα, μπορέσουμε να βρούμε και άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε για να απαντήσω σε όλα όσα δέθηκαν σήμερα. Και επίση, ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε, δημερώσουμε στη διάθεσή σα. Ευχαριστώ ιδιαίτερω για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για το ότι μας διαθέσατε το χρόνο σας που μας δώσατε τις πληροφορίες και για το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. <coughs> Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε με τις ε, ψηφοφορίες. Φαντάζομαι ότι θα έχετε όλοι σας, ε, όλη την κάρτα σας. Gut. Können wir beginnen, meine Damen Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η ημερήσια διάταξή μα έχει κατά τη τροποποιηθεί. Πάντω είμαστε μέσα στο χρόνο μα. Ψηφίζουμε λοιπόν για το ε, θέμα των μεθόδων πρόσβαση στην κυβερνητική υπηρεσία, η οποία προσφέρεται από το Παγκόσμιο Σύμβουλο Δορυφορική Ραδιοπλοήγηση που προέκυψε από το πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Σημείο 9 τη ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε λοιπόν. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 23. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΑφΕ 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΑφΕ 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά Εγκρίνεται. Αποχέ τις ξέχασα, λέει ο πρόεδρο. 26 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. άφετε 15, 16 λέει ο πρόεδρο. Υπέρ, κατά, Αποχέ. Ε, εγκρίνεται. άφετε 17 υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Αφετ 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα λοιπόν η ΑΦΕΤ 20, από την ΑΦΕΤ 20, 20, 22, 23, 24, 23 και 6. Για αυτά ψηφίζουμε ε, ενσώματι όλα Ψηφίστηκαν. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άφετ 25 ε, ως προστίκη, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άφετ 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άφετ 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άφετ 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα... Α, εσείς μπορείτε να τα έχετε ψηφίσει όλα μαζί. Μα εγώ δεν είπα ακόμα να ψηφίσουμε. Πάμε τώρα στην 29. Λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετε 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30... Άφε 32 μπερδεύτηκε πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 33 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 32 με προφορική τροποποίηση του αντέλφου κυρίου Λάμπερς που δεν χρειάζεται να τη διαβάσει, υπέρ παρακαλώ κατά αποχές ε, επίσης εγκρίνεται. Πάμε στο παράρτημα 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφετ 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές αποχές απορρίπτεται. Άφετε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 ως προστίκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άφε 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, αφετ 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 σκέτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 ε, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10, αφετ 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αφετ 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 22, 22 με προφορική τροπολογία του Σαντέλφου Λάμπερτς υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 12 συνάδελφου Λάμπερτς πάλι προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, αυτή τη φορά απορρίπτεται 13 παρακαλώ υπερκατά. κατά Μισό λεπτό, τι θέλετε να ελέγξουμε στο 12, μα ήταν σαφές. Ελέγχουμε, με βάση περιπτώσει. Ας ελέγξουμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποια στιγμή τη μηχανή. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ο ένας, ένας από το ΕΛΚ ε, περισσεύει, μία ψήφο στο ΕΛΚ παραπάνω, έκλεισε λοιπόν και το αποτέλεσμα είναι ε, οριακά απορρίφθηκε. Πολύ αριακά. Πολύ καλό αυτό που κάνετε, που ζητήσατε ε, να το ελέγξουμε. Ποιος το έκανε, ποιος το ζήτησε παρακαλώ, να τον βραβεύσω. 13 λοιπόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αφέτε 7, 7 είχε πει 17 πρώτης και κάνει λάθος, 7 ήταν υπέρ κατά αποχές. Ε, και τώρα τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Μπορούμε να αρχίσουμε να ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πάλι ένας ε, περισσεύει μία ψήφος από το ΕΛΚ. Περισσεύει μία ψήφος από το ΕΛΚ. Έκλεισε. Πολύ ωραία. Τώρα το λόγο θα λάβει ο κύριος Γκλάντ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τους σκιώδης ηγητές ε, για την καλή συνεργασία και κυρίω για το πνεύμα ε, συμβιβασμού. Και νομίζω ότι αυτό το πνεύμα σύναψης συμβιβασμών που υπήρξε αυτή τη φορά, αν εξακολουθήσει να υπάρχει και στις τριμερείς θα τα καταφέρουμε μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά και για τη δουλειά και για τις συμφορίες. Ρεκόρ πετύχαμε σήμερα, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, στο υπαριθμόν 10 ε, για την ευρωπαϊκή ευρυζωνικότητα. Η κυρία Τζαβέλα είναι η συγκητριά μας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν θέλετε να συζητήσετε, να εγκαταλείψετε την αίθουσα γρήγορα, με ταχύτητα ή ε, τουλάχιστον να μιλάτε σιγά, να μην ακούγεστε. Η κυρία Τζαβέλα παρακαλώ έχει το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. The aim of this... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να παρουσιάσει μια καλά ισορροπημένη έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των κρατών μελών και προκειμένου να δώσει επίσης κίνητρα για τους Ευρωπαίους ε, πολίτες και τους καταναλωτές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, Το 2003 η Επιτροπή είπε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα πια για όλους τους πολίτες μας. Η ευρυζωνικότητα συνεπώς συμπεριλαμβάνεται. Τον Ιούλιο του 2010 στην ε, Φιλανδία έγινε νομικό δικαίωμα η ευρωζενικότητα, διότι βοηθάει την εκπαίδευση και η νομοθεσία λέει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα τουλάχιστον σε ένα μεγαμπιτ ε, σύνδεση ευρυζενικότητας. Έτσι λοιπόν από την αρχή του 2011 στην Ισπανία όλοι οι πάροχοι ενθαρρύνονται να προσφέρουν καλές τιμές για την ευρυζωνικότητα. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε μεταξύ μας. Προσπαθώ να πω ότι το 2013 πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στην ευρυζενικότητα, να υπάρχουν ελάχιστοι στόχοι για τις αγροτικές περιοχές, τουλάχιστον 2 ΜΜ για τους χρήστες και 24 στις αστικές περιοχές. Έτσι όπως αναφέρει και η έκθεση. Όμως, βάσει των στόχων του 2020, εγώ υπογραμμίζω ότι προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους για την ευρυζωνικότητα το 2020, η ψηφιακή ατζέντα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους ενδιάμεσα για το 2015, για το 2018 και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε εθνικό επίπεδο. Έπειτα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα εδώ είναι εκείνα της χρηματοδότησης. Το 2011 η κρατική ενίσχυση ήταν 1,8 δις ευρώ, ρεκόρ. Και πάνω από 100 σε εφόσον φτάσουμε, σημαίνει 200 με 300 δισεκατομμύρια ευρώ ότι χρειάζεται χρηματοδότηση. Και 38 με 58 δις για να πετύχουμε το 100% κάλυψη ευρυζωνικότητας με 30 Mbit το 2020. 80% όσων χρησιμοποιούν νέες υποδομές πολιτικού μηχανικού Πρέπει να βρούμε λοιπόν νέες καινοτόμε μεθόδους χρηματοδότησης αυτού του τεράστιου σχεδίου. Για παράδειγμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ρόλο που παίζουν οι εταιρικέ σχέσεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα, να δούμε τι μπορεί να γίνει με τη χρηματοδότηση και να στοχεύσουμε την βελτίωση ε, απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό θα γίνει εφόσον συνεργαστούμε καλά μεταξύ μας. Και όσο συνεχίζεται η συζήτηση για το ομόλογα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω ότι η ευρυζωνικότητα είναι ένα καλό ε, πρόγραμμα υποδομών, το οποίο θα μπορέσει έτσι να χρηματοδοτωθεί από τέτοια ε, προγράμματα ομόλογα. Μην ξεχνάμε ότι 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την σύνδεση, αλλά βρισκόμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες χώρες όπως είναι η Κορέα ή η Ιαπωνία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να θυμόμαστε ότι μιλάμε για διαφορετικές αγορές και ίσως δεν είναι καλό να κάνουμε τέτοιου είδους συγκρίσει. Πάντω, για να έχουμε μια αποτελεσματική οικονομική ανάπτυξη στην ευρυζενικότητα, πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανάπτυξη των βασικών ε, υποδομών στα σχολεία, σε επιχειρήσεις, σε διάφορα επίπεδα κυβέρνηση, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα παράδειγμα. Τι κάνει η Ρουμανία πρόσφατα για την σύνδεση με τα νοικοκυριά δεν έχει την κατάλληλη υποδομή. Έχει επενδύσει πάρα πολύ για τα νοικοκυριά και χρησιμοποιεί την μέθοδο της οπτικής ίνας σε κεραίες ε, τηλεφωνίας και φροντίζοντας ε, να ε, βρει και τα χρήματα για να φτιάξει υποδομές κάτω από το έδαφος. Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολύ ακόμα, όμως θα ήθελα εδώ να ακούσω τους συναδέρφους τι έχουν να πούνε. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, πριν ολοκληρώσω, θέλω να κλείσω με το εξή. Με δύο ακόμα ζητήματα. Πρώτον, όλες οι προσπάθειές μας όσον αφορά το ρόλο της ευρυζωνικότητας θα χαθούν εφόσον στις προτεραιότητές μας δεν συμπεριλάβουμε στρατηγική για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δεύτερον, αναγνωρίζω ότι οι υποχρώσεις μας για τις ε, καθολικές υπηρεσίες πρέπει να συμπεριλάβουν και αυτή την υπόθεση. Και ο λόγος για τον οποίο δεν τον αναφέρω εδώ στην έκθεσή μου είναι ότι θα υπάρξει ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τα τέλα, τέλη Μαΐου ή το αργότερο αρχές Ιουνίου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα στην άλλη έκθεση. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάντως πολύ για την προσοχή σας και προσδοκώ σε συνεργασία με τους, στοιχειο... με τους σκιώδεις εισηγητές. Σίγουρα στο τέλος θα έχουμε μια καλά ισορροπημένη έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, οκτώ έχουν ζητήσει το λόγο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε όλοι σας να μιλήσετε κατά το μέγιστο δύο λεπτά. Κυρία Βαλιάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τζαβέλα για μια ε, ισορροπημένη έκθεση θα έλεγα. Αναφέρεται όλες τις ε, αρχές, ε, την υποδομή, ε, τις υποδομές για τον ανταγωνισμό, την μη διακριτική μεταχείριση, τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών, την τεχνολογία, όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Επίσης, εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι η συγγήτρια τελικά αναφέρθηκε και στην κρατική βοήθεια στην έκθεση. Όμως, Θέλω να πω το εξή. Στην περίπτωση αυτή η ανακοίνωση τη Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ακριβή όσον αφορά τι κρατικέ επιδοτήσει και ε, είναι λίγο περίεργο το ότι αυτό δεν αναφέρεται στην έκθεση. Βέβαια, εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει για να μην υπάρχει και συνταγωνισμού, αλλά σε απομακρυσμένε περιοχέ ίσω εκεί θα πρέπει να υπάρχει κρατική ενίσχυση. Και δεύτερον, η πολιτική με στόχους. Αυτό μοιάζει να είναι ε, χαρακτηριστικό της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής και ίσως να μην πολύ αρέσει, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να φέρονται οι στόχοι που συμφωνήθηκαν για την ψηφιακή ατζέντα. Η ευρυζωνικότητα να ε, υπάρξει σε όλους τους Ευρωπαίους μέχρι το 2013 και το 25% των οικοκυριών συνδεδεμένα με διαδίκτυο. Αυτό θα μπορούσε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα για να στηριχθούν τα μέτρα της αγοράς. Ε, ίσως λοιπόν θα κάνω τροπολογία ε, στο εδάφιό σας το C για να αναφερθεί αυτό που σας είπα. Όσον αφορά την παράγραφο υπαριθμών 29. Δεν μπορώ να στηρίξω τη σύσταση task force ομάδας κρούση όπως προτείνετε εσείς. Και δεν θέλω να συσταθούν ε, νέα γραφειοκρατικά εργαλεία. Και δεν αναφέρεται και αυτή η task force για ποιο λόγο να συσταθεί. Δεν είναι σαφές. Δεν βλέπω την υπεραξία σύστασης μιας τέτοιας ομάδας και επιπλέον αυτή θα κατακυριαρχείται από μεγάλους παίκτες και έτσι θα υπάρξει διακριτική μεταχείριση και στρέβλωση ανταγωνισμού. Τέλος, το cyber security στην παράγραφο 3. Αυτό μου αρέσει και ενισχύει ε, την τροπολογία μας γιατί ε, εμείς ε, θέλουμε ως στόχο να υπάρχουν ψηφιακοί, ε, λεωφορείο, ψηφιακές, ψηφιακοί διάδρομοι ένα, μικρό έλλειμμα, αυτό που είπατε για τη Ρουμανία κύριε Τζαβέλα. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία και θέλω να πω, ελπίζω ότι οι επενδύσεις της Ρουμανίας ε, στην ευρυζωνικότητα αυτά δεν μπορούν να αποτελούν κριτήριο για αποτελέσματα οικονομικής ανάπτυξης γιατί αυτό θα ήταν πράγματι πολύ φτωχό παράδειγμα και το αποτέλεσμα, το γεγονός μάλλον το θέμα των ινών, των οπτικών ινών. Αν δείτε λιγάκι στις πόλεις μας και όλους αυτούς τους πυλώνες με τα καλώδια υπάρχει κανονισμός που ζητάει από τις επιχειρήσεις να τοποθετήσουν υπόγεια τα καλώδια αυτά. Άρα ούτε και αυτό το παράδειγμα είναι καλό. Συνάδελφος Κάλφιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την εισηγητρία την κυρία Τζαβέλα για την εξαιρετική έκθεση που υπέβαλε και για το πολύ ανοιχτό πνεύμα και την ευθεία με την οποία ετοίμασε την έκθεση αυτή. Να σταθώ σε ορισμένα σημεία που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να συμπληρώσει κάπως το όλο πνεύμα της έκθεσης. Πρώτα απ' όλα, κάτι που ήδη αναφέρθηκε για την ουδετερότητα του δικτύου και την παροχή καθολικών ε, υπηρεσιών. Όταν μιλάμε για την ε, πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα, θα μπορούσαμε να θεωρούμε ότι αυτή η υπηρεσία είναι καθολική, εφόσον πρέπει να παρέχεται ως ισότιμο δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους πολίτες. Έπειτα, οι εξελίξεις στον τομέα πληροφορίας, επικοινωνίας και τεχνολογιών. Για το cloud computing που λέγαμε και χθες και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις θα συσχετιστούν οπωσδήποτε με το τι θα γίνει και στην ευρυζωνικότητα και τη διαχείρισή της. Στηρίζω λοιπόν ε, θερμός αυτό που λέει η, η συγγήτρια για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο για αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και για άλλα θέματα που θα πρέπει να μας οδηγήσουν να διαμορφώσουμε μια συνολική στρατηγική ασφάλειας. Τώρα σε αντίθεση με την ε, συνάδελφο από την Άλντε, Συμφωνώ με την ιδέα να δημιουργηθεί μια ομάδα δράση που να συζητήσει και να προσπαθήσει να διαμορφώσει το μέλλον τη ευρυζωνικότητα στην Ευρώπη. Και θα πρέπει εκεί να συμπεριληφθούν οι ε, ενδιαφερόμενοι, όχι μόνο μεγάλες εταιρείε, αλλά ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκπρόσωποι των καταναλωτών, η ΕΝΗΣΑ και άλλοι οργανισμοί και φορείς, ώστε να έχουμε μεγάλη εκπροσώπηση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων και να διαμορφώσουμε έτσι τις εξελίξεις στην ευρυζωνικότητα. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση και με το πώς θα ιεραρχήσουμε τα διάφορα κονδύλια. Νομίζω ότι πρώτον πρέπει να στηρίξουμε την ευρυζωνικότητα με ε, ε, ιδιωτικά κονδύλια αλλά και τα δημόσια. Τα κρατικά θα είναι πολύ σημαντικά διότι ούτε το ένα μπορεί να λειτουργήσει κατά το 100% ούτε το άλλο. Και βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τη διάσταση των περιφοριών κατά την υλοποίηση του προγράμματο Ευχαριστούμε ο κύριο Χέκμαρκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει η ασφάλεια, η ηλεκτρονική ασφάλεια, γιατί ε, αυτό παίζει ρόλο, έχει σημασία για το ρόλο που θα διερματίσει το διαδίκτυο. Κάτι άλλο, το έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν και μου αρέσουν όλα αυτά που αναφέρονται, αλλά κατά κάποιον τρόπο αισθάνομαι ότι πρέπει να έχουμε ακόμα πιο υψηλέ ε, φιλοδοξίε. Εξώσον, και μάλλον κατανοώ την εισηγήτρια, γιατί βεβαίω είναι πολύ εύκολο να αναφέρει κανεί υψηπετεί στόχου, ε, χωρί όμω ε, να υπάρχει καμία ελπίδα να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Παρ' αυτά όμω πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπο σκέψη μα. Γιατί αν δεν είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε το βέλτιστο με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ε, θα παρέμβουν άλλοι. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής απόφασης, είναι και θέμα σύστασης του σωστού πλαίσιου επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να παραμείνουμε εστιασμένοι στο να ανοιχτούμε σε όσο δυνατόν μεγαλύτερες ε, εμπορικές ε, επενδύσεις. Γιατί βλέπουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρχει ταχεία διάδοση της ευρυζωνικότητας. Βέβαια αυτό είναι και παράδοξο, διότι από τη στιγμή που ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι και θέμα φορολογούμενο, αυτομάτως προκύπτει και ένα όριο ε, στον τομέα αυτό. Και όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Αρκεί να δει κανεί ε, τους προπολογισμούς των κρατών μελών κατά την επόμενη δεκαετία. Ε, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί όσον αφορά τις επενδύσεις Γι' αυτό λοιπόν λέω να προβούμε σε ιδιωτικές επενδύσεις. Παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για κρατική βοήθεια. Γιατί δεν υπάρχει αυτή ας πούμε σε άλλους τομείς όπου δεν υπάρχουν εξελίξεις. Πάντως για να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα και αποτελεσματικότητα ε, Εκεί σας λέω θα μπορούσαν να υπάρξουν ιδιωτικέ επενδύσεις για να επεκταθούμε όχι μόνο γεωγραφικά αλλά όσον αφορά και το δυναμικό, τον όγκο. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει να παραμείνουμε στοχευμένοι και να γνωρίζουμε ότι ε, τα ενία θα τα έχουν ιδιώτες επενδυτές και μετά θα ακολουθούμε εμείς με τις κρατικές ενισχύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα εναντίον πολιτικών στόχων, έτσι όπως δηλώνονται εδώ. Δηλαδή, κατά της αύξησης της ταχύτητας ή ε, κατά το ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρύτερου κύκλους πολιτών. Αλλά το θέμα της ουδετερότητας. Στο σημείο α αναφέρονται πολλές εναλλακτικέ λύσεις για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ευρυζωνικότητα. Για το χαλκό, για τα καλώδια, για χωρίς καλώδιο, δορυφορικά κτλ. Ενώ στο σημείο 9, εκεί που μιλάμε για το ψηφιακό μέρισμα, μιλάμε για τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις. Θα έπρεπε εδώ να υπάρχει μία εξαίρεση και αυτή να είναι δορυφόρη. Γιατί αν δούμε τι μπορούν να κάνουν οι δορυφόροι είναι η δυνατότητα μετάβασης του σήματος από απόσταση. Δεν έχουμε άλλη τέτοια λύση. Οι δορυφόροι μπορούν να λύσουν αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα οι συχνότητες να προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές και ώστε να χρησιμοποιούνται οι φορείς αυτή η τεχνολογική ικανοποιητικά και απρόσκοπτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζέις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η ευρυζωνικότητα, η ταχεία δηλαδή πρόσβαση στο διαδίκτυο πολλά μπορεί να προσφέρει όπως και η οικονομική ανάκαμψη. Εδώ Θυμόμαστε τι αλλαγές έφερε η επανάσταση του ηλεκτρισμού στα τέλη του 19ου αιώνα. Εδώ λοιπόν οι νέε επενδύσεις για την ανταγωνιστικότητα και μέσω και της κρατικής στήριξης είναι η καλύτερη δυνατή εγγύηση για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει μέχρι το 2020. Για το θέμα αυτό ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Θεωρώ πρωταρχικής σημασίας ως την ανταγωνιστικότητα, την ελεύθερη ανταγωνιστικότητα την ε, πρόσβαση όλων των πολιτών στα νέα δίκτυα. Για να έχουμε βιώσιμο ανταγωνισμό θα μπορούσαμε να ευνοήσουμε συγκεκριμένες υποδομές και βεβαίως να δούμε κατά πόσον εδώ μπορεί να αξιοποιηθούν κρατικές βοήθειες. Να μην υπάρξει μονοπόλιο στην αγορά. Δεύτερο ζήτημα. Σκόπιμο θα ήταν τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα δίκτυα όλων των ε, φορέων που εμπορεύονται τις οπτικές αυτές ίνες. Θα μπορούσαμε έτσι να επιτρέψουμε την πραγματική χειροπιαστή περικοπή του κόστους για τις υποδομές, επιτρέποντας και σε άλλα μερίδια της αγοράς να αναπτυχθούν και φροντίζοντας να έχουμε πολλαπλασιαστική, ε, κέρδη πολλαπλασιαστικά από την, ε, από την καλωδίωση. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να προσαρμοστούμε με τρόπο λογικό ώστε και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να απολαμβάνουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές αλλά με συγκατημένο κόστος. Θα πρέπει λοιπόν έτσι το τιμολόγιο να υπολογίζεται βάσει του συνολικού κόστου, ακόμη και του εμέσου. Και θα πρέπει να προβλέψουμε αρχές υπολογισμού και σε επίπεδο κρατών μελών, για να μπορέσουμε να περάσουμε με τρόπο πιο ισότιμο στην ευρεία διάδοση της ευρυζωνικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε ιδιαίτερα στη συνάδελφο Τζαβέλα για την εξαιρετική σύνταξη τη έκθεση και τη συστήνουμε ακριβώς τη. της Αυτέ τι αλλαγές προκειμένου να βελτιωθεί η παρουσία της ανταγωνιστικότητας στην αγορά του συγκεκριμένου ζήτηματο και να προστατευτούν περισσότεροι Ευρωπαίοι καταναλωτέ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφο Τσίκαου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Τζαβέλα για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Θεωρώ ότι είναι καθοριστική σημασία να υποστηρίξουμε εδώ τις υπάρχουσες υποδομές για να μπορέσουν να καλύψουν και το ψηφιακό περιεχόμενο. Το 2008 είχαμε ήδη ένα πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα εκατομμύριο ευρώ ότι θα αποδοθούν ως κονδύλιο για την κάλυψη του αναγκών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός δεν επετεύθηκε και τελικά δεν εκταμιεύτηκε το σχετικό κονδύλιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε θέσει ένα στόχο που πρέπει να επιτευχθεί στο τέλος του 2013. Δεν θα είναι δυνατό κάτι τέτοιο εάν δεν προβλεφθεί το ανάλογο κονδύλιο από τον προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πρέπει να δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στις απομακρυσμένες περιοχές, στις απομονωμένες και αραιοκατοικημένες οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν έχουν αναγκαστικά πρόσβαση στο διαδίκτυο, ούτε θέλουν αναγκαστικά να προβλέψουν ε, υποδομέ για τέτοιες περιοχές. Ε, οι εταιρείε ειδικά σκέφτονται και το κέρδος σε αυτές τις περιπτώσεις. Να γιατί χρειάζονται και κρατικά κονδύλια προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες υποδομές και για τις απομονωμένες αεροκατοικημένες περιοχές. Να καλυφθούν και αυτές. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να σχολιάσω είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κυβερνοασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν νομίζω καλή ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει μια έκθεση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το εξετάζει το θέμα αυτό, ας υπάρξει έστω μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία από τη δική μα Επιτροπή για το θέμα. Όλοι οι μηχανισμοί προστασία στην κοινωνία τη πληροφορία είναι ιδιαίτερης ε, σημασίες. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι φορείς της κοινωνίας της πληροφορίας γνωρίζουν επαρκώς τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους. Και εδώ μιλάμε και για τους παρέχοντες και για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους εκείνους ε, οι οποίοι στήριξαν ανεπιφύλακτα την εισηγήτρια και την επένεσαν επίσης. Σύμφωνα και εγώ. Πρόκειται για μια πολύ καλή ισορροπημένη έκθεση ε, που στρέφει κυρίως την προσοχή της στο που ακριβώς χρειαζόμαστε κίνητρα. Ε, χρειαζόμαστε κυρίως ε, από ιδιώτες επενδυτές ε, για να προάγουμε την ευρυζωνικότητα και επίσης αναφέρεται και στην έκθεση που καλείται το κράτος να παρεμβαίνει για να διασφαλίσει την ευρυζωνικότητα σε όλους. Δύο σύντομες παρατηρήσεις θα μου επιτρέψετε. Πρώτον, θεωρώ ότι στην έκθεση πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο το ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Εδώ καλούνται οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να εντοπίσουν που υπάρχουν κενά στην αγορά, ε, που δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, που πρέπει να παρέμβει το κράτος ε, για να συσταθεί υποδομή ευρυζωνικότητας. Και νομίζω, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει να εντοπίσουμε ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ο ρόλος του Ευρωπαίου εισαγωγικά ε, ρυθμιστή, ε, ποιος είναι ο ρόλος του οργανισμού ΕΝΙΖΑ, πώς μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταθέσουμε ε, συστάσεις. Νομίζω ότι αν το κάνουμε αυτό θα είναι ακόμα καλύτερη έκθεση. Και ένα πράγμα που δεν υπάρχει είναι το θέμα της δορυφορικής επικοινωνίας. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια προσθήκη στην έκθεση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορεί μπορεί κανεί την ευρυζωνικότητα να την εγγυηθεί και με τη χρήση τη δορυφορική επικοινωνία, με χαμηλό κόστο. Αυτό μπορείτε να το προσθέσετε. Και κάτι άλλο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θυμάμαι στη συζήτηση πριν από δύο χρόνια για το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Τότε αναφέρθηκε επανειλημμένα ότι ε, για την ευρυζωνικότητα και την υποδομή τη. αυτό ε, που είναι πολύ δαπανηρό είναι το να μεταφέρονται οι συνδέσει και να υπάρχει η καλωδίηση, η τοποθέτηση των καλωδίων. Αποφασίσαμε Βλέπουμε λοιπόν τότε ότι όποτε πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο σε κάποιο κράτος δηλαδή να τοποθετούνται οι αγωγοί και τα καλώδια, αυτομάτως να γίνεται και πρόβλεψη για τοποθέτηση μελλοντικά οπτικών ινών για την ευρυζωνικότητα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό συνέβη σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, ίσως η συγγήτρια μπορεί να μας πει κάτι, μήπως το ξέρει γιατί αν αυτό είναι το πρόβλημα, το roll-out δηλαδή των καλωδίων, η τοποθέτηση είπα εγώ με πρόβλεψη για οπτικές ίνες, ε, θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα κρατημέλη. Υπάρχει κάποια πρόοδος. Η κυρία Ντελκαστήγιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να συγχαρώ τη συναδελφό μας ε, κυρία Τζαβέλα διότι η πρότασή της είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να υπενθυμίσω τη συζήτηση που είχαμε όταν είχαμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την υπόθεση αυτή. Υπήρχε μια συνένεση σχετικά με το ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει όχι μόνο αυτή την υπόθεση για την ευρωζενικότητα, αλλά και την σύσταση που είχε ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσβαση στα δίκτυα, όπως επίσης και την υπόθεση για το ραδιοφάσμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για λόγους που εξήγησε και ο συγκητής κ. Χόρτμακ, η έκθεση αυτή, και ό,τι έχει να κάνει με την ευρυζωνικότητα, να είναι στην ίδια κατάσταση. Επιμένω δηλαδή για το ότι τα 800 να είναι έτοιμα για το 2013, αλλά επίσης να υπάρχει και επέκταση για τα 700 Mbps, όπως αναφέρεται και στην έκθεση για το διαφάσμα, στην πρόταση τη σχετική. Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συνοχή. Και για άλλους λόγους, τους οποίους δεν θέλω να επιμείνω τώρα, και άλλες φορές, σε άλλη συζήτηση, έχουμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει την δυνατότητα αυτή η ευρυζωνικότητας. Άρα λοιπόν θέλουμε να προωθήσουμε έναν ανταγωνιστικό τομέα. Από την άλλη, και θέλω να συγχαρώ ε, από αυτού την κυρία Τζαβέλα, έχει εισαγάγει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ρύθμισης. Κάτι πολύ σημαντικό ως προσανατολισμός στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς για ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό ρόλος που μπορεί να παίξει ένας τέτοιος οργανισμός Ευρωπαίων ρυθμιστών. Μπορεί να υποβάλω κάποια τροπολογία από αυτού. Είναι πολύ σημαντικό, επιμένω, να υπάρχει συνοχή στην άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό, σύμφωνα με την θεωρία αυτή ότι υπάρχει ένα πακέτο που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ραδιοφάσμα και να συμπεριλάβουμε και εδώ τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια αποστολή, έτσι όπως έχει στην έκθεση για το ραδιολεκτρικό φάσμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι διπλά ενδιαφέρουσα. Απ' τη μια βλέπουμε ότι χρειάζονται νέα δίκτυα μεγαλύτερης χωρητικότητας για να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη μεριά πρόκειται για μια αναγκαιότητα για τους πολίτες μας. Μιλήσαμε για την χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε πρόκειται για την εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όμως πώς μπορούμε να οθήσουμε τους διάφορους φορείς να χρηματοδοτήσουν σε τομείς που είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί. Έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται ε, καλύτερη πρόσβαση. Έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι εναλλακτικέ λύσεις. Έχουμε ήδη παραδείγματα προγραμμάτων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή χάρη στα μέσα που αναφέρει η συγκήτρια. Επίσης, θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους τους πολίτες η ταχύτητα. Είναι και θέμα καινοτομίας και θέμα οικονομίας, άρα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση όλων των πολιτών στο διαδίκτυο. Στα πλαίσια της συζήτησης που είχαμε για την οδηγία για τη δυσυνοριακή υγεία, επέμεινε εγώ πάρα πολύ για την εξαποστάσεως ιατρική. Δυστυχώς, δεν οδήγησε σε κάτι στο κείμενο, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη ήταν επιφυλεκτικά. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε αυτό το τομέα. Γιατί και αυτό είναι θέμα οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την Επιτροπή ο κύριος Μάτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως σας είπα και κατά την τελευταία συνεδρίαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χαιρετίζει την έκθεση αυτή. Ε, συνεργαστήκαμε στενά με την εισηγήτρια και πάρα πολύ καλά. Από τα πολλά σχόλια που έγιναν, εγώ δεν θέλω τώρα να σπαταλίσω το χρόνο σας αναφερόμενο σε όλα αυτά, αλλά θα κάνω κάποιες γενικής φύσεως παρατηρήσεις. Καταρχήν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τονίσω και εγώ, πως και άλλοι, το ε, τι θα κάνουμε με αυτή την έκθεση. Η βάση της ε, στρατηγικής ε, του 2020 ε, έχει ως στόχο η στρατηγική αυτή την δημιουργία της συνεργασίας. Αναφέρθηκαν επίσης πολύ στην ανταγωνιστικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη. Οι πληροφορίες, οι τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να συμβάλλουν κατά το ίμιση στην αύξηση της παραγωγικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο κίνητρο. Γι' αυτό ασχολούμεθα με αυτό το θέμα. Και ως εκ τούτου ε, η έκθεση αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική. Εμείς ε, καταθέσαμε προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο του πακέτου ευρυζωνικότητας και τώρα νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε και πέρα από αυτό. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ θετική ε, και υπάρχουν πολλά στοιχεία που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Αρκετοί σχολίασαν το, τη δυνατότητα να περιοριστεί το κόστος της επένδυσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει, όπως ε, ανέφεραν και άλλοι, ότι οι ιδιωτικέ επενδύσεις είναι ένας καθοριστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Οι επενδύσεις αυτές ίσως να μην υπάρχουν σε όλους τους τομείς, αλλά όπως είπε και η συγγήτρια, Μιλάμε για περίπου 250 δις ευρώ απαραίτητα για να επιτευχθούν οι στόχοι. Και αυτά θα έρθουν σε μεγάλο βαθμό από τον ιδιωτικό τομέα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε το κόστος αυτής της επένδυσης. Και αναφέρθηκαν και ορισμένα άλλα πράγματα αναφέρθηκε παραδείγματο χάρη ε, το πώ τοποθετούνται οι ίνες ε, ε, όταν γίνονται παράλληλα και άλλα έργα, αυτό που λένε Αμερικανοί, ω στρατική dig wants. Εμείς εκείνο που προτιθέμεθα να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με κράτη-μέλη, να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα κράτη-μέλη ήρθαν σε εμά εκφράζοντα την επιθυμία να συνεργαστούμε καλύτερα για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και στις 23 ε, Μαρτίου θα έχουμε μια συνάντηση με τα κράτη-μέλη όπου θα προσπαθήσουμε όλα αυτά που σας είπα να τα προωθήσουμε. Αυτό που υπογραμμίσαμε είναι ότι όλα τα κρατημέλη πρέπει να έχουν μια στρατηγική προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι με μονομένα κρατημέλη θα μπορέσουν να επιτύχουν τους ευρωπαϊκούς στόχους. Πρέπει να υπάρχει κάποια εναλλαγή σε αυτά και πρέπει να συνεργαστούμε. Και τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Σύντομα θα αναφερθώ ε, στους δορυφόρους που το, τους έφτιαξαν αρκετοί. Από την άποψη της Κομισιόν εμείς από πλευράς ε, νομοθεσίας πρέπει να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι. Εάν οι δορυφόροι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους, πολύ καλά θα είναι μέρος της στρατηγικής. Αλλά εξ όσων γνωρίζω, ακόμα οι δορυφόροι τεχνολογικά δεν είναι σε θέση ε, να προσφέρουν το στόχο 30 MB. Επίσης, ε, εξ όσων γνωρίζω, οι δορυφόροι μπορούν να, να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ε, με ε, πρόσβαση ε, χωρίς καλωδίωση. Ασύρματη. Εμείς λοιπόν μιλήσαμε με τους ε, ε, χειριστές των δορυφόρων και θα συνεχίσουμε να συζητάμε για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκε λοιπόν η ασφάλεια από αρκετούς και πράγματι εμείς συμφωνούμε με όλους όσοι υπογραμμίζουν τη σημασία της ασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται παράλληλα με άλλα θέματα της ψηφιακής ατζέντα και γι' αυτό δεν επαναλαμβάνεται εδώ. Όμως θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους ότι η ασφάλεια είναι το κλειδί των μελλοντικών μας πράξεων και ενεργειών. Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν. Κλείνω ευχαριστώντας την κυρία Τζαβέλα για μια πολύ χρήσιμη και θετική έκθεση. Κυρία Τζαβέλα, θέλετε εσείς να λάβετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον κύριο Μάθερν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά μαζί. Αγαπητοί συνάδελφοι, στην Επιτροπή αυτή είχαμε μία γενικότερη έκθεση, την έκθεση Καστίλιο, για την ψηφιακή ατζέντα. Επίσης, είχαμε και την έκθεση του κ. Χόρκμαν για τα ραδιοφάσματα. Συνεπώς, αυτό που προσπαθώ να κάνω με αυτή την έκθεση είναι να κρατήσω μια συνοχή και με την ψηφιακή ατζέντα και με την έκθεση του κύριου Χόρκμαν. Ελπίζω να τα κατάφερα. Τα σχόλιά σας τα σημείωσα, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε συνάντηση με τους γιώδεις εισηγητές πριν την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών που είναι 23 Μαρτίου. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ρωτάω την γραμματεία γι' αυτό. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών. 23 Μαρτίου. Δύο σχόλια παρακαλώ όμως έχω να κάνω εδώ. Ένα πράγμα που σχολιάσατε πολύ είναι το θέμα της Task Force. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει την σύνθεση και την λειτουργία μιας Digital Assembly. Νομίζω λοιπόν ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να συμπεριλάβουμε την Task Force και πρέπει να έχουμε όλους τους ε, εταίρους εκεί. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια αγορά η οποία αναπτύσσεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Πρέπει λοιπόν να έχουμε εδώ και την αγορά και τους καταναλωτές. Δεύτερο, το σχόλιο του κύριου Χόρκμαν για τις κρατικές ενισχύσεις. Και για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ε, σωστό το σχολείο. Η πρότασή του είναι πολύ καλή, πιστεύω. Συμφωνώ. Κυρία Νίμπλερ, δεν γνωρίζω τι γίνεται στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα έργα αυτά. Θα μπορούσε ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει σε αυτό. Συνεπώς, θα συναντηθούμε οι σκιώδεις εισηγητές και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 23 Μαρτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ε, Γραμματεία για την βοηθειά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Αν δεν επιθυμεί κανείς άλλος να ζητήσει το λόγο, μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η κυρία Τζαβέλα ήδη μας ε, επισήμανε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάσταση είναι 23η Μαρτίου και 25-26 Μαΐου θα γίνει η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ θερμότατα και πάμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Εφόσον βέβαια είναι εδώ η συνάδελφος από την Επιτροπή Προεπολογισμών. Χρειαζόμαστε την κυρία Μπαλτσάνη. What can we do now? The Basini is not there? Are you news about? No. If you want, I can call the Barzani, Francesca. Yeah, we, we called her office. Yeah, and? Nobody there. Eigentlich müsste die Kollegin Balsini jetzt hier sein, aber... Κανονικά θα έπρεπε να εδώ η κυρία ε, Μπαλτσάνη. Εμείς προσπαθήσαμε να την πάρουμε τηλέφωνο και στο γραφείο. Ψυχή δεν υπάρχει. Ίσως να έρχεται εδώ. Ίσως να είναι καθοδόν. Αυτό βρίσκω ως ε, έξυπνη εξήγηση. Ούτε και μπορούμε να ξεκινήσουμε και με το άλλο <laughs> θέμα της μήνυσης διάταξης. Λείπουν και εκεί οι συνάδελφοι. Αλλιώς θα πήγαινα στο ε, μεθεπόμενο. Ας περιμένουμε λιγάκι. Εντάξει. Έτσι καλώς τι να κάνουμε. Gut, dann darf ich äh, in Ihrer aller Namen die Kollegin Balsini ganz herzlich begrüßen. Sie ist Καλωσορίζω λοιπόν τη συνάδελφο κυρία Μπαλτσάνη, η οποία είναι αρμόδια για τον ε, Γενική Συγκήτρια για τον Προεπλισμό του 2012 και η κυρία Μπαλτσάνη μας έστειλε μια επιστολή ε, και μας πρότεινε να συζητήσουμε ε, σε βάθος ε, για τα βασικά θέματα. Αυτό το βρήκαμε καλή ιδέα και αποφασίσαμε να κάνουμε τώρα μια συζήτηση, όχι ανταλλαγή επιστολών. Γι' αυτό λοιπόν σας καλωσορίζω θερμά, χαίρομαι που είστε εδώ. Και ίσως θα ήθελα να σας δώσω εσάς το λόγο. Στην αρχή έχουμε μισή ώρα για αυτό το θέμα της μηνυσίας διάταξης στη διάθεσή μας. Ίσως μπορείτε εσείς ε, ε, να τοποθετείτε και μετά ε, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους για τη συνάντηση που οργανώσατε. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκομαι σήμερα εδώ είναι πολύ απλός. Εδώ θέλουμε να έχουμε άμεση συμμετοχή σα και να σα παρουσιάσουμε τι ειδικέ συνθήκε που ισχύουν για τη διαδικασία αναθεώρηση του προπολογισμού. Η διαδικασία του προπολογισμού, όπω ξέρετε, είναι μακρά, περίπλοκη και ανακαλύψαμε ότι με τη θέση στην, σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο περίπλοκα από ό,τι απλούστερα οι ε, διαθεσμικέ σχέσει μεταξύ των αρχών του προπολογισμού γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αναγκαίο και περισσότερο και αποσκόπιμο ευθύ εξ αρχή ε, από τη διαδικασία αυτή και τη στιγμή που ξεκινάει ε, στην Επιτροπή Προπολογισμών να παρακολουθούμε τι γίνεται και στι υπόλοιπε ειδικέ επιτροπέ. Και αυτό για έναν καθοριστική σημασία στατηγικό λόγο. Επειδή βρισκόμαστε σε στιγμές οικονομικών δεσχεριών, όπως αυτές που τώρα ζούμε, έτσι θα πρέπει αμέσως να έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Και λέγοντας προτεραιότητες εννοώ όχι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, αλλά τη ίδια της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυτό είναι στατηγική σημασία. Διότι σημαίνει ότι αμέσως θα κάνουμε τις σωστές επιλογές Η πρότασή μου την οποία θα έχετε μπορέσει να δείτε είτε στο έγγραφο εργασία, το πρώτο έγγραφο που πρότεινα, είτε στο σχέδιο ψηφίσματο που πρόκειται να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή η πρόταση είναι πρόταση ισχυρή, ώστε να καθορίσουμε τις προτεραιότητες των διάφορων τομέων για τον προπολογισμό του 2012 στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής του 2020. Νομίζω ότι η ανάγκη ε, ε, ανανέωσης που προέκυψε και από τον περσινή χρονιά, να έχουμε ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση και επιβεβαιώθηκε φέτος με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για πρώτη φορά, είναι μια πράξη ε, ε, πραγματικού συντονισμού των ε, κρατικών εθνικών προπολογισμών προ την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού. Έτσι, μπορεί σε 10 χρόνια να επιδιώξουμε και να πετύχουμε ε, του στόχου τη στρατηγική του 2020. Θα πρέπει ήδη λειτουργικά να εξυπηρετήσουμε την επίτευξη των στόχων αυτών. Μιλάμε για στόχου που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσε πράξει, ε, τι οποίε έχουμε εγκρίνει, την εγκρίναμε μόλι την τελευταία στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου, να επιβεβαιώσουμε λοιπόν ότι οι στόχοι αυτοί για μα είναι πρώτη τη σημασίας. Και εδώ ε, οι προτεραιότητες αυτές αγγίζουν ακριβώς τις αρμοδιότητες της Επιτροπής της συγκεκριμένης. Όχι γιατί στην ε, στατική του 2020 αναφέρονται οι επενδύσεις, αλλά και η έρευνα, η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που θα προέρχεται από μια Ευρώπη ανταγωνιστικότερη στη διεθνή της διάσταση. Αυτό λοιπόν που αμέσως πρότεινα στα πλαίσια της Επιτροπής Προπολογισμών ήταν να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία περί προπολογισμού και να ανοίξει για τις επιτροπές τις ειδικότερε ό,τι αφορά τις θέσεις των προτεραιοτήτων των τομεακών προτεραιότητε που στη συνέχεια θα γίνουν όχι μόνο αναπόσπαστο τμήμα τη δική μα ερμηνεία του ψηφίσματο μετά την πρόταση τη Επιτροπής τη 20 η Απριλίου, όπου εκεί σκοπεύω να κάνω κάποιε προτάσει για τι αρχέ Μαΐου, αλλά και για να έχουμε ευθύ εξ αρχή ένα συγκεκριμένο εργαλείο, για να μπορούμε με τρόπο διαφανή, συνεπή και ξεκάθαρο να δούμε ποιε είναι οι τροπολογίε που θα πρέπει να κάνουμε σε συγκεκριμένα σημεία του προπολογισμού. Ε, έτσι θα τεθούν συγκεκριμένες πολιτικές σαφείς προτεραιότητες. Το θέμα προτεραιότητας για το οποίο σας καλώ ήδη να αρχίσετε, να σκέφτεστε για την ερχόμενη περίοδο του προπολογισμού είναι ε, δύο όψεων. Πρώτα απ' όλα ότι έχουμε θετικές προτεραιότητες. τι θέλουμε δηλαδή να συμπεριλάβουμε ως προτεραιότητα για τον προπολογισμό του 2012 και τι είναι αρνητική προτεραιότητα. Τι θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να το στηρίξουμε όπως το παρελθόν. Αυτό βεβαίως σημαίνει συνολικά ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε πρώτα απ' όλα πριν από οποιαδήποτε άλλη επιλογή για την ερχόμενη περίοδο του προπολογισμού. Αυτή η εξέταση αφορά και τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις τα, πολιτικά, τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις δεν έρχονται να προσθεθούν στο προπολογισμό, απλώς παίρνουν ένα μέρος του υπάρχοντος περιθωρίου. Περιορισμένο μερίδιο σε σχέση και με το γενικότερο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών. Σε σχέση λοιπόν με όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει ευθύ εξ αρχή να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε ποιε είναι οι προθέσεις τη κάθε μια ειδική επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη. Έτσι, όσο των δυνατόν νωρίτερα, οπωσδήποτε πριν το καλοκαίρι, θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια προσωρινή ε, ένα προσωρινό κατάλογο προτεραιοτήτων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έπειτα σε μια σκόπιμη κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, προτεραιότητες για ανάγνωση και ερμηνεία της πρότασης προπολογισμού που θα γίνει 20, στις 20 Απριλίου, μια ε, εξέταση όρημη και συνειδητή, ώστε μετά να κάνουμε και χρησιμοποιημένε αριθμητικέ προτάσει. Αποτελεσματικέ. Και πριν το καλοκαίρι να έχουμε καταλάβει ποια πολιτικά προγράμματα και ποια, πιλωτικά μάλλον και ποιε προπαρασκευαστικέ δράσει πρέπει να συνεχιστούν τα περιθώρια, το είπα και προηγουμένω, είναι περιορισμένα. Αυτό ε, το ξέρουμε γιατί βρισκόμαστε και σε αυτή τη φάση περίοδο προγραμματισμού. Αλλά επίση να θυμίσω ότι η πτυχή αυτή για τα περιορισμένα περιθώρια φέτο μπορεί να μα οδηγήσει και σε πιο χειροπιαστή συγκεκριμένη χρήση της ευελιξίας του 5% που διαθέτουμε από το άρθρο 137 της Διαθεσμική Συμφωνίας. Έτσι μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό το θέμα, ε, διότι τώρα το λόγο ουσιαστικά τον έχετε εσείς. Εσείς πρέπει να συμμετάσχετε σε αυτή τη φάση. Εγώ σας έδωσα μια γενική κατεύθυνση, ένα γενικό προσανατολισμό. Πρέπει αμέσως να διαλέξουμε μεταξύ των γραμμών του προπολογισμού που θεωρούνται σημαντικέ και σχετίζονται με τη στρατηγική του 2020 και τι θερμοδιότητε αυτέ τι επιτροπέ. Και έπειτα, κατά την κρίση σα, την πείρα σα και τι θεωρίε σα, πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να ενισχυθεί ή τι να περιοριστεί εν ώψη του μελλοντικού προπολογισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, και πράγματι σωστά επισημάνατε ότι σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό ε, πρέπει να είμαστε σαφέστεροι, να μιλάμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Γιατί, Γιατί τα κονδύλια, τα διαθέσιμα θα είναι περιορισμένα. Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μας προσφέρθηκε να συζητήσουμε. Καταρχήν, συνάλφος Πιτικόφα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, κυρία Μπαλτσάνη, να σας ευχαριστήσω θερμά ε, για το ότι ήρθατε σήμερα εδώ ε, για να γίνει αυτή η συζήτηση με την Επιτροπή μας. Πέρυσι η συγγήτρια, η κυρία Χέρτσοκ, ε, από κοινού με εσάς, κύριε Πρόεδρε, συνέταξε μία επιστολή όπου συμφωνήθηκαν οι προτεραιότητες της Επιτροπής. Ε, συμφωνήθηκαν προτεραιότητε από κοινό με τους συντονιστέ. Θεωρώ λοιπόν ότι η Γενική Εισηγήτρια θα συμπεριλάβει τα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και συζήτηση με τους ε, συντονιστές για το ε, κατά πόσον μετά τη συζήτηση μας το λάβει η χώρα εδώ θέλουμε να συντάξουμε μια επιστολή. Καταρχήν λοιπόν να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το σημείο βάρους που προβάλλεται κυρία Μπαλτσάνη στο έγγραφό σας. Λέτε δηλαδή ότι είναι απαραίτητο η δημοσιονομική πολιτική να προσαρμοστεί προς τη στρατηγική για το 2020, στρατηγική 2020. Και οι εμβληματικές πρωτοβουλίες και οι στόχοι αφορούν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα για τα οποία είμαστε εμεί αρμόδιοι. Άρα δηλαδή πρέπει να υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στους στόχους της στρατηγικής και τη χρηματοδότηση σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι η Επιτροπή αυτή, όλα αυτά που σας είπα, τα θεωρεί μεγάλη προτεραιότητα. Πράγματι λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευτούμε στην πράξη το ευρωπαϊκό εξάμεινο για να επιτύχουμε καλύτερο συντονισμό. Και όπως και εσείς ε, και εγώ θεωρώ ότι απορρέει μεγαλύτερη θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη χρήση ευρωπαϊκών επενδύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την πράσινη τεχνολογία. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ε, συνεργαστούμε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε το εξής. Η ε, προσέγγιση αυτή που έχει σχέση με τα headline goals και τα flagship initiatives, αυτά ε, δεν πρέπει να περιστούν, του αντίον να επεκταθούν περαιτέρω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τα εξετάσουμε όλα αυτά και σε σχέση ε, με το εξάμεινο που θα ακολουθήσει. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική συμμετοχή. Εσείς είπατε ότι πρόκειται να κάνει η Επιτροπή σας. Ίσως λοιπόν κύριε Πρόεδρε εμείς ως Επιτροπή Ήτρε ε, μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για θέματα που μας αφορούν. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Περνάω στη δεύτερη. Πέρυσι κυρία, ήδη, ήδη είδαμε, βιώσαμε ότι η κυρία Χέρτσοκ ε, ένα σημαντικό τμήμα της δουλειάς της το αφιέρωσε στη χρηματοδότηση ε, μεγάλων προγραμμάτων, προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Και είδε ότι αυτή η χρηματοδότηση έρχεται σε σύγκρουση με χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο υπαριθμών 7. Τότε λοιπόν, πέρυσι, είπαμε με την κυρία Χέρτσο και φέτος πρέπει να ξαναπούμε ότι ένας καθοριστικός στόχος αυτής της Επιτροπής είναι να εμποδίσουμε η χρηματοδότηση των προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας να έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, σε ε, άλλα προγράμματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7. Ε, τρίτη παρατήρηση. Στον τομέα της ενέργειας Εκεί πρέπει να, δώσουμε, να ρίξουμε το βάρος μας. Παραδείγματο χάρη, η χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση για τους στόχους SET. Εκεί λοιπόν ε, δεν θα πρέπει να ε, μπούμε απαραίτητα στη συζήτηση περί ενέργειας. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνουμε αυτό για να επισημάνουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενεργειακή ασφάλεια και μια πολιτική ενέργειας διαρκείας η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της, της ε, την κλιματική αλλαγή και τις κλιματικές προκλήσεις. Ε, είναι σημαντικά όλα αυτά και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Επιτροπή μας. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή μας, εμείς ε, και το ΙΤΕΡ η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος ΙΤΕΡ, η χρηματοδότηση του προγράμματος δεν θα πρέπει να οδηγήσει ε, σε αρνητικές επιπτώσεις σε άλλα παρεμφερή προγράμματα. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Κατά την άποψή μου αυτό που είναι σωστό ε, θα ήταν να έχουμε ξεχωριστό προπολογισμό για το πρόγραμμα Γκαλιλαίο και να καθορίσουμε ποια είναι τα ποσά εκείνα του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία στο μέλλον θα διατίθενται για το πρόγραμμα Γκαλιλαίο και ποια περισσεύουν. Και ό,τι περισσεύει, μάλλον πώς το πρόγραμμα Γκαλιλαίο θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο και από εκεί και πέρα μπαίνουν τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούν και οι χρήστες. Όσον αφορά τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο για το ΣΥΠ όσο και για το πρόγραμμα πλαίσιο ε, πρέπει να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και συντονισμός της αναθεώρησης του προγράμματος με την στρατηγική 2020. Αυτό που επίσης με ενδιαφέρει είναι η χρηματοδότηση για Risk Sharing Facility, για το μέσο εκείνο που επιτρέπει τον επιμερισμό των κινδύνων. Ε, μου είπαν ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μέσο, εργαλείο και γι' αυτό λοιπόν εγώ λέω ότι τα κονδύλια για το εργαλείο αυτό θα πρέπει να αυξηθούν. Και τέλος, με την ευκαιρία της έκθεσης της κυρίας Τζαβέλα, Ακούσαμε και αυτό το περίφημο όρο ψηφιακή Ευρώπη. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν νέα κονδύλια χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την χρηματοδότηση υποδομών ευρυζωνικότητας. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να θίξουμε και ένα άλλο φλέγον θέμα της παρούσας ε, κατάστασης περιβιομηχανίας το θέμα της ε, αποτελεσματικότητας των πόρων. Αυτό είναι ένα θέμα ε, με μεγάλη προτεραιότητα. Και τέλος, όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις preparatory actions, τις προκαταρκτικές ενέργειες, έχουμε ακόμα λίγο καιρό στη διάθεσή μας, αλλά εγώ θα έλεγα και καλό να το πούνε αυτό και τους ε, σκιώδης και την εισηγήτρια. Όλοι μας λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε αυτά τα ε, προαναφερθέντα θέματα έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να καταθέσουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Ο συνάδελφος κύριος, ή, ή συνάδελφος με συγχωρείτε, κυρία Χέρτσοκ. Ευχαριστώ πολύ. Μια που συζητάει ήτρε για τον προπολογισμό, Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Παλτζάνη. Είναι η πρώτη φορά που η συγγύητής από την Επιτροπή Προπολογισμών έρχεται εδώ σε εμά. Και αυτό αποδεικνύει ότι ο προπολογισμό τώρα με τη διαδικασία της συναπόφασης αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολόκληρο. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία, να την πω έτσι, μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτρεπών, πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό νέο. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο Βουτικόφερ δείχνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλά. Αυτό δείχνει προς το παρόν και ελπίζω ότι όντως έτσι θα γίνει όπως έγινε και πέρυσι. Συμφωνώ πάντως με την κυρία Παλτζάνη απόλυτα για το ότι το 2012 είναι το έτος που μας οδηγεί μέχρι το 2020. Δεν πρέπει να περιμένουμε το 2019 για να θυμηθούμε τότε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για το 2020. Όχι. Κάθε χρόνο πρέπει να φροντίζουμε να προχωράμε έτσι ώστε να πλησιάζουμε όλο και περισσότερο το στόχο μας για το 2020. Και εντάξει, ξέρουμε ότι η θέση του Συμβουλίου είναι δεν υπάρχουν χρήματα για τα επόμενα δύο χρόνια στις δημοσιονομικές προοπτικές. Πρέπει όμως να βρούμε τρόπους ώστε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τα ήδη υπάρχοντα χρήματα, για τους στόχους εκείνους δηλαδή που πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας, για αυτούς τους σκοπούς. Και ξέρουμε ότι μία από τις δυσκολίες μας προέρχεται από, την, ναι, από τις νέες αρμοδιότητες της συνθήκης της Λισαβόνας, καινοτομία, τουρισμός κλπ, το οποίο δεν είναι στην Επιτροπή μας και είναι εντελώ καινούργια πράγματα τώρα. Περισσότερα από αυτά είναι αρμοδιότητα της δικιάς μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και γι' αυτό εμείς υποφέρουμε περισσότερο να δούμε πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό. Πάντως θέλω να πω ε, ευχαριστώ στην Επιτροπή Προπολογισμών για την εξαίρετη συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας. Όντως ε, ήρθαν στη δικιά μας τη γραμμή πέρυσι και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε κρατώντας την ίδια γραμμή και φέτο. Πιο συγκεκριμένα τώρα για κάποια ζητήματα. Οι πρωτοβουλίε αποτελούν προτεραιότητα όχι μόνο για μας στην Ήτρα, το Flexifar, αλλά είναι και σημαντικά πράγματα για τους περισσότερους Ευρωπαίους. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, πρέπει να δείξουμε ότι προχωράμε προς την κατεύθυνση που θέλουν. Και η ενεργειακή ε, αποδοτικότητα και όλα τα, τα, τα θέματα που καίνε τους πολίτες θα χρηματοδοτούνται παρκώς. Ήδη πέρυσι είχαμε μια δυσκολία. Τα χρήματα δηλαδή που πηγαίνανε στην ανταγωνιστικότητα και όχι μόνο και διάφορες διοικητικές γραμμές αντιμετώπισαν δυσκολίες στο Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε εμείς ως Επιτροπήτρε ότι οι γραμμές που έχουν να κάνουν με την δίκηση είναι εξίσου σημαντικές όσο και τα χρήματα που πηγαίνουν σε άλλες γραμμές σίγουρα τέθηκε σε αντιπαράθεση το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με τα μεγάλα προγράμματα. Όμως το Γαλιλαίο, το πρόγραμμα αυτό, είναι πολύ σημαντικό και άλλα. Η στρατοχική για τις τεχνολογίες επίσης και άρα πρέπει να φροντίσουμε να χειριστούμε αυτά τα θέματα διαφορετικά. Να βρούμε δηλαδή μια λύση για το συνολικό κόστος. Ενώ όλα τα μεγάλα προγράμματα τώρα υποφέρουν. Συγχρόνως πρέπει να διασφαλίσει η Επιτροπή μας τη συνέχιση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνήθως το πρόβλημα σε αυτές είναι το αντίθετο, ότι είναι πολύ μικρές, υπερβολικά μικρές σε σχέση με άλλα θέματα που απορροφούν κονδύλια από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Είναι πολύ σημαντικό πάντως το πώς βλέπει τις αρμοδιότητες της Ήτρε η εισηγήτρια και την ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών είσαστε ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο, οπότε σίγουρα ό,τι αποφασίσουμε μαζί θα περάσει και στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Κάντριον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σε ευχαριστώ Φραντσέσκα και για την ε, δική σου την ε, εισήγηση και παρέμβαση που ε, είναι κατά την άποψή μου η καλύτερη που μπορούσε να υπάρχει και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να μιλάμε για μια βέλτιστη διαδικασία, ε, για έναν καλύτερο συντονισμό. Αυτό είναι κάτι που ε, σίγουρα μας ε, δίνει κίνητρα, αλλά δεν φτάνει. Στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα γκρίναμε την κοινοβουλευτική πρωτοβουλία που αφορούσε ακριβώς αυτές τις νέες μορφές χρηματοδότησης. Και εδώ πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στα ευρωομόλογα από τα project ομόλογα, project bonds. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, βέβαια η αρχή είναι ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν ε, τα ευρωμόλογα με βάση τις συνθήκες αλλά αυτό των ε, project bonds είναι ένα θέμα που νομίζω ότι χάνεται σιγά σιγά. Πάντως εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω για να ξέρουμε και εμείς τι είδους προτάσεις θα σου κάνουμε ας δούμε το τι ακριβώς εξελίσσεται και ας δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα. Γιατί εγώ νομίζω με τον κανονικό προπολογισμό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε ε, κάτι πραγματικά σημαντικό ε, σε σχέση με την στρατηγική του 2020. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε σημαντικά κίνητρα για να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Για να είμαστε λοιπόν φιλόδοξοι και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίσιμη οικονομική στιγμή, οικονομική συγκυρία στην Ευρώπη σω Ίσως αυτό που θα μπορούσαμε να βρούμε είναι η λογική των ΣΔΙΤ. Ευχαριστώ κυρία Μπαλτζάνη για τις ε, νέες αυτές ιδέες ότι αφορά τη γενικότερη συζήτηση για τον προπολογισμό του 2020. Το κοινοβούλιο μα έχει εργαστεί πανηλημμένω για την επεξεργασία προπολογισμών και καταλαβαίνω ότι πάντοτε υπάρχουν πρωτοβουλίε που υποβάλλουν οι βουλευτέ και μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευρείε. Προσπαθούμε να είμαστε λοιπόν εδώ ανοιχτοί στο πνεύμα και να σκεφτούμε ποιε είναι οι κυρίε προθέσει των διαφόρων κρατών, γενικότερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι χρειάζονται πολύ περισσότερα κονδύλια. Νομίζω ήδη σήμερα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ποιε θα είναι οι στρατηγικέ μα προτεραιότητε και στόχοι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Τι θέλουν να χρηματοδοτήσουν για το 2012. Για να μπορέσουν να στοχεύσουν καλύτερα και την εμβέλεια των δικών μας των προτάσεων. Όπως εδώ υπόθηκε, πρέπει να έχουμε υπόψη ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης που διαθέτουμε. Το Συμβούλιο θα πρέπει ενδεχομένως να υποβάλει και ιδέες για τέτοιες καινούργιες πηγές. Ξέρουμε ότι έχουμε το Ταμείο των Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι ιδιωτικέ επενδύσει, τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Κάποιοι μηχανισμοί στο παρελθόν δεν έχουν λειτουργήσει επαρκώ. Ιδίω όταν μιλούμε για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περίπου 15 δι από τα ευρωπαϊκά κονδύλια παρέμειναν στους λογαριασμούς αχρησιμοποιητά. Πολλά είναι αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Η στατηγική που προτείνεται, η στατική του 2020, μπορεί να φέρει κάποιες αλλαγές. Δεδομένων και όλα των πρόσφατων εξελίξεων στην Ιαπωνία. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξεύρει κάποιες προτεραιότητες για το 2012 είτε ε, προβλέψουμε νέα προγράμματα, είτε απλώς προωθήσουμε τα υπάρχοντα. Η κυρία Εκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που ήρθε ως εδώ και για τις προτεραιότητες που ανέφερε. Εγώ μιλώ εκ μέρους όχι μόνο ε, των εισηγητών, αλλά και ως υπεύθυνη για τη στρατηγική του 2020. Όταν οι πολιτικές ομάδες εξέτασαν το θέμα τη στρατηγικής αυτή και το ψήφισμα ε, περί συγκεκριμένου θέματο πέρσι και φέτο. είδαμε ότι υπάρχουν κάποιε ασυνέμειες μεταξύ των στόχων που θέλουμε να πετύχουμε και το τι προβλέπει σχετικά ο προπολογισμό. Είναι λοιπόν πολύ συγκεκριμένη δουλειά που πρέπει να γίνει. Να πάμε σε διάφορε γραμμέ του προπολογισμού και να είμαστε βέβαιοι ότι ε, στοχεύουν πολύ συγκεκριμένα στη βιώσιμη ανάπτυξη που έχουμε εγκρίνει με ευρία πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι εύκολη δουλειά, είναι όμω εξαιρετική σημασία. Πολύ με ανησυχεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ιδίω από δύο οπτικές γωνίες. Πρώτα απ' όλα, επειδή και στην ανακοίνωση για το κλίμα διαβάσαμε κάποια στοιχεία, όχι τόσο για το κλίμα αυτό καθεαυτό, αλλά για τις επενδύσεις. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις φτάνουν στο 19% του ΑΕΠ μας. Οι κεφαλουχικές επενδύσεις. 19%. Η Κίνα 48% η Ινδία 35%, η Κορέα 26%. Προκειμένου λοιπόν να πετύχουμε τους στόχους του 2020 πρέπει να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις. Η έρευνα και η καινοτομία βεβαίως είναι ένα σημαντικό στοιχείο, η ενέργεια και οι υποδομές της επίσης. Όμως γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η τιμή της ενέργειας πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον και ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία λόγω ε, έλλειψη πόρων. Η Ιαπωνία δεν τα έχει πάει και πολύ καλύτερα όπω βλέπουμε. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και των Ευρωπαίων πολιτών είναι να προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Εάν δούμε και διεθνώς τι συμβαίνει ως προς τις επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία. Και πάλι σε χαμηλά επίπεδα βρισκόμαστε σε σχέση με τις Ηνωμένες Εάν κοιτάξετε του Ευρωπαϊκού αριθμού και του αντιπαραβάλλεται με του Αμερικανικού, θα δείτε ότι τα κρατικά κονδύλια είναι τα ίδια περίπου, όμω, αν δούμε τι ιδιωτικές επενδύσει, χανόμαστε, χανόμαστε στο πέλαγος τη ανταγωνιστικότητα. Δεν μιλάμε για μικρή απόσταση εδώ, μιλάμε για τεράστιε αποστάσει. και εδώ μην ξεχνάμε και την Κίνα. Οι επενδύσει λοιπόν στην ε, έρευνα και την ανάπτυξη και την καινοτομία είναι σημαντικέ. Το ίδιο και η στοχοθέτηση για την στατική του 2020. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αξιοποιούνται όσα ήδη διαθέτουμε. Και το ΣΕΤ, ε, το ε, πρόγραμμα ΣΕΤ για την ε, στατηγική έρευνα ενέργεια και τεχνολογία. Το αναφέρει διαρκώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν δούμε τη χρηματοδότηση, είναι λιγότερο από 50%. Και ένα μέρο είναι από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, αλλά και σε χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να το δούμε. Τι θα γίνει αν αποσύρουν κονδύλια σε κρίσιμε στιγμέ. Το θέμα είναι λοιπόν τι θέλουμε να παραμένει στο πρόγραμμα, τι θέλουμε να ε, λειτουργήσει. Γιατί δεν θα συμβούν όλα αυτά χωρί χρηματοδότηση. Είναι τεράστιο το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το τέταρτο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Από συνταγματική κιόλα άποψη, νομίζω ότι μα ανησυχεί ιδιαίτερα οι αποφάσει για το ΙΤΕΡ λαμβάνονται από έναν μόνο φορέα και η χρηματοδότηση καταβάλλεται από και διασφαλίζεται από άλλον. Αυτό το θα πρέπει να το φροντίσουμε. Σε όλε τι περιπτώσει, όποιοι λαμβάνουν τι αποφάσει θα πρέπει να διασφαλίζουν και τη χρηματοδότηση. Και μάλιστα, σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοσιονομική πειθαρχία του προγράμματο ITER, βλέπετε πολλά να υπονομεύονται. Από τη μια οι τιμέ, από την άλλη έλλειψη συνέπεια για την ιεράρχηση τη πειθαρχία και τη χρηματοδότηση. Εδώ λοιπόν νομίζω το κοινοβούλιο δεν είναι ο πιο δύσκολο μιλήσει στην όλη συζήτηση. Μάλλον το Συμβούλιο είναι, έχει αυτό το ρόλο. Επειδή λοιπόν θα περάσετε στι διαπραγματεύσει, σα εκλυπαρώ. Ζητήστε του να κρατήσουν επιτέλου τι υποσχέσει του, να παραμείνουν πιστοί σε όσα δεσμεύτηκαν να κάνουν, ιδίω σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δύο ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Να είστε πολύ σύντομοι, παρακαλώ. Αλλιώς η κυρία Μπαλτζάνη δεν θα έχει χρόνο στη διάθεσή της για να σας απαντήσει. Ο κύριος Διάντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Φραντσέσκα. Πραγματικά ήταν πολύ επικοδομητική η πρωτοβουλία και η συζήτηση που είχαμε. Ιδίω η συμμετοχή των διάφορων ειδικών επιτροπών είναι σημαντικό να γίνει αυτή η συζήτηση για τον προπολογισμό, για τη διαδικασία του προπολογισμού την ίδια. Έχουμε όλοι καταλάβει ποιες είναι οι συνέπειες της κρίσης. Οι πόροι δεν είναι πλέον ε, ανεξάρτητοι. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε ορθώς αυτούς τους λίγους πόρους που υπάρχουν. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα που τίθεται και εδώ πραγματικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Η ποιότητα των δαπανών όχι μόνο η ποσότητα. Μας ενδιαφέρει κυρίως η ποιότητα. Ποιότητα της δαπάνης, ιδίως ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Επενδύσεις οι οποίες είναι... πρέπει να είναι παραγωγικές. Ιδίως στην περίοδο της ανάπτυξη που πρέπει να στοχεύουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, τη θέση εργασίας. Αυτά είναι τα βασικά θέματα που τουλάχιστον εγώ τα βρίσκω πρώτη τη σημασία. Επίση, πρέπει να εντοπίσουμε και να δώσω έμφαση σε κάποια στοιχεία τη παρουσίασή σου, δηλαδή τι προτεραιότητε, τι στρατηγικέ μα επιλογέ. Για τι προτεραιότητε ακριβώ. Κατά πρώτον πρέπει να έχουμε έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να στοχεύσουμε πρώτα απ' όλα σε αυτά τα δύο στοιχεία. Δεν θα υπάρξει ανα... Αν δεν υπάρξει μάλλον ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει μέλλον. Αν δεν επενδύσουμε στην έρευνα και την καινοτομία, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Αυτό είναι ο πρώτο στόχο. Δεύτερο ζήτημα που τίθεται. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε κατά το βέλτιστο τρόπο και πώς θα παροτρύνουμε τις ε, χρηματοδοτήσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι στο παραγωγικό οικονομικό πεδίο της Ευρώπης καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές χρειάζονται εργαλεία αλλά και στόχους που να είναι επικεντρωμένες στις ανάγκες τους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Πώς να βοηθήσουμε λόγω χάρη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κάνουν έρευνα. Και κλείνω, τελείωσα ήδη, η ενέργεια. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα σήμερα είναι ιδιαίτερη επικαιρότητα, ιδίω μετά τα όσα συνέβησαν στην Ιαπωνία. Νομίζω ότι οι επενδύσει προ αυτή την κατεύθυνση αξίζουν, ιδίω αυτή τη φάση, ιδιαίτερη προσοχή και μέσα στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Σε κάθε τήσιο προπολογισμό, ένα μέρος των προγραμμάτων συγχρωματοδοτείται από τον προπολογισμό των κρατών μελών και των ε, τοπικών αυτοδικήσεων επίσης. Ε, θέλω και αυτό να το πω. Συνεπώς, αυτό που λείπει σήμερα είναι η σταθερότητα των δημοσιονομικών των χωρών μελών. Και αυτό υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να μειωθεί ο δημόσιος προπολογισμό, ο κρατικός, που έχει σαν συνέπεια τη μείωση του προπολογισμού και των ε, διαφόρων αυτοδικήσεων. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει αρκετή συγχρηματοδότηση είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να μην μπορέσει να καλυφθεί ούτε ο ευρωπαϊκός προπολογισμό γιατί θα αποσυρθούν οι τοπικές αυτοδιοίκησει από τα διάφορα προγράμματα. Και έχουμε τέτοιε πληροφορίες. Μπορεί δηλαδή τελικά να αποδειχτεί ότι οι αρχές που υιοθετήθηκαν για τον προπολογισμό του 2012 συνδέονται με την στρατηγική μας και οι αρχές αυτές θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Εσείς τι λέτε. Άλλη ερώτηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέρος των κονδυλίων αυτών όλο και μικρότερο βέβαια για την καινοτομία ή για άλλους στόχους. Οι μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις χρειάζονται πιστώσεις. Με κάποια κριτήρια βέβαια δίνονται οι πιστώσεις αυτές και συχνά τελικά οι τράπεζες δεν δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις πιστώσεις που χρειάζονται και γι' αυτό αποσύρονται από ορισμένα προγράμματα που κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα θετικά, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζω λοιπόν ότι υπάρχει αυτός ο σημαντικός κίνδυνος σήμερα, κίνδυνος που έχει να κάνει με τον προπολογισμό του 2012 και κυρίως με τις βασικές αρχές αυτού του προπολογισμού. Κύριε Μπαλζάνη θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε όσο μπορείτε στις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έγιναν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε όλες οι παρεμβάσεις. Όχι απλώς ενδιαφέρουσες, αλλά και πολύ χρήσιμες χρήσιμες ακριβώς από την οπτική γωνία ενό εντοπισμού των προτεραιοτήτων που πρέπει συγκεκριμένα να συμπεριληφθούν στον προπολογισμό το 2012. Μου φαίνεται λοιπόν πολύ σημαντική η προσπάθεια που πρέπει να αρχίσει αμέσως να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες ε, για την στρατηγική του 2020. Θα πρέπει λοιπόν αυτή να προσαρμοστεί και να καλύψει τις προτεραιότητες αυτής της Επιτροπής. Μιλήσαμε για έρευνα, καινοτομία και ενέργεια. Για μια νέα προσπάθεια, έντονη προσπάθεια να αναζητήσουμε ασφαλή ενέργεια, ανανεώσιμη ενέργεια. Ε, είναι τόσες πολλές οι προτεραιότητές μας ε, υπό την οπτική της στρατηγικής του 2020 που μπορούμε να τις αποφασίσουμε και να τις στηρίξουμε ήδη από την Επιτροπή αυτή. Αλλά και κάτι άλλο προέκυψε από τη συζήτηση και είναι ενδιαφέρον γιατί ίσω για πρώτη φορά ε, μετά από τι διάφορε συζητήσει που είχαμε τι ειδικέ επιτροπέ ακούγεται το θέμα τη χρηματοδότηση ε, συνεχώ. Ε, το είπαν πολλοί συνάδελφοι και για την ψηφοφορία που είχαμε στο Στρασβούργο σε σχέση με την έκθεση Ποδηματά. Εδώ είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσον όλοι υποφέρουμε από την ανεπάρκεια πόρων που πλήττει τον προπολογισμό μας εδώ. Δεν ζητά μόνο η Ευρώπη περισσότερες παρεμβάσεις, όλοι ζητούν περισσότερη Ευρώπη. Αυτό το θεωρώ πολύ θετική εξέλιξη. Είναι όμως και δύσκολο να καλύψουμε νέες αρμοδιότητες που έχουν προκύψει και αυτό είναι ένα πρόβλημα αξιοπιστίας θεσμικής. Διότι Θέλουμε να αυξηθούν οι αρμοδιότητες, αλλά πρέπει να έχουμε και τα μέσα να τους δώσουμε ένα συγκεκριμένο μέλλον και να έχουμε κύρος και αξιοπιστία θεσμική. Είναι λοιπόν σημαντικό, δεν μπορεί να τα καθορίσει αυτά ο προπολογισμός μόνος του. εμείς θα τα αποφασίσουμε και να θυμίσω το εξή. Πέρσι η όλη διαδικασία του προπολογισμού ε, αναγκάστηκε να συμπεριλάβει και άλλα ζητήματα, όπω οι δημοσιονομικέ προοπτικέ συζητιόνταν ταυτόχρονα. Έγινε πιο δύσκολη η όλη διαδικασία ώστε να κλείσει το πρώτο σχέδιο του προπολογισμού και η πρόβλεψή του. Εδώ λοιπόν, κατά τρόπο συγκεκριμένο και ρεαλιστικό, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ο στόχο μα θα επιδιωχθεί σωστά. Δηλαδή να ορίσουμε ένα προπολογισμό για το 2012 όσο το δυνατόν καλύτερο, αλλά εφικτό, δυνατό. Πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστέ. Τα θέματα που τέθηκαν, τα, οι μελλοντικοί πόροι, τα ομόλογα είναι σημαντικά και από, άλλη πολιτική, και από άλλη οπτική γωνία στα πλαίσια τη πολιτική μα συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε, διότι θα πάρουμε κάποιε πολιτικέ αποφάσει στα πλαίσια του προπολογισμού. Η λύση που θα εξεύρουμε την προσεχή εβδομάδα στην Ολομέλεια της, των Βρυξελών θα καλύπτει και αυτά τα θέματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε πολιτικά ανοίγματα. Πώ μπορούμε να μεταφράσουμε συγκεκριμένε πρωτοβουλίε σε αυτή τη φάση σε προκειμένου στη συνέχεια να έχουμε και αριθμητικά στοιχεία και προτάσει που τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και επίση να συνοδεύσουμε όλε αυτέ τις προτάσει με πολιτικά έγγραφα ώστε να δώσουμε μια ισχυρή όθηση και σε σχέση με τα όσα αποφασίστηκαν στο Στρασβούργο. Έπειτα υπάρχει και το θέμα τη συγχρηματοδότηση. Συγχρηματοδότηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει αρνητικό αντίκτυπο για τι επιλογέ που κάνουμε στον προπολογισμό. Διότι ακριβώ η έλλειψη πόρων των δημόσιων αρχών και θυμίσετε εδώ και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Η έλλειψη λοιπόν, η ανεπάρκεια που γνωρίζει ο κοινωνικός, οικονομικός και θεσμικός ιστός κάνει σχεδόν ε, μάταιες τις προσπάθειες προπολογισμού που κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λείπουν οι σχέσεις συνεργασίας. Αυτό είναι ένα θέμα που ε, προκύπτει ξανά και ξανά. Και αυτό γιατί έχει να κάνει με την αξιολόγηση της ε, βαρύτητας που διαθέτει ο καθένα στα πλαίσια τη διαδικασία ε, προπολογισμού. Πρέπει να ενισχύσουμε την οικονομική συνεργασία και τα σημεία επαφή ε, του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού με τα εθνικά κέντρα. Όχι μόνο για οικονομικέ συνεργασίε, αλλά για να ξεπεράσουμε και φραγμού. Φραγμού λόγου χάρη τη έλλειψη χρηματοδότηση και τη έλλειψη ισορροπία μεταξύ πόρων που αυτή τη στιγμή θέλουμε να συμπεριλάβουμε στον προπολογισμό μα και πόρου που θα μπορούσαν να δαπανηθούν επειδή δεν υπάρχουν αρκετέ δυνατότητε χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι απαραίτητο να έχουμε την ε, ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των κρατών μελών, ώστε και εκείνοι να συνειδητοποιήσουν ότι γι' αυτό μα χρησιμεύσε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Για να καταλάβουμε πολύ συγκεκριμένα σε τι είναι απαραίτητο να επενδύσουμε, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μπορέσουμε να αποφεληθούμε πλήρω από τι δυνατότητε που δημιουργούνται με τον κοινοτικό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Άρα, Α αρχίσουμε να εργαζόμαστε αμέσω για τον προπολογισμό τη Ένωση. Να είναι σαφή αυτό ο προπολογισμό. Να υπάρχει και ένα μήνυμα για του επιμέρου εθνικού προπολογισμού και οι αρχές τους να σκεφτούν εκείνες πώς θα εκτελέσουν τις οικονομικές τους επιλογές. Έτσι, αυτές οι ίδιες οι επιλογές θα είναι συνεπείς με τις δικές μας και θα μπορέσουμε να μειώσουμε, γιατί δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τελείως τα προβλήματα, θα μειώσουμε τα προβλήματα σε χρηματοδότηση. Έτσι, τα επιμέρους κράτη-μέλη θα καταλάβουν ότι ο ε, ευρωπαϊκός προπολογισμός τους δίνει κάποιους γενικούς προσανατολισμούς που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και κάποιε ευκαιρίε από την ε, θέση αυτή. Έτσι λοιπόν αμέσω να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη να συμπεριληφθούν αυτέ οι προτεραιότητε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προπολογισμού ώστε να επηρεάσουμε και του εθνικού. Να αναζητήσουμε επικοινωνία με το τι συμβαίνει στα εθνικά μέσω των βουλευτών. Επίση ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ποιότητα των δαπανών. Το έθεσε ο συνάδελφο Ντεάντζελη. Η ποιότητα λοιπόν των δαπανών, η οποία προφανώς πρέπει να εξεταστεί είναι θέμα προτεραιότητας. Αλλά πρέπει να το δούμε με τρόπο επικοδομητικό. Όχι αρνητικά. Να θέσουμε κάποιε προτεραιότητες, ε, θε, εξετάζοντας όπου είναι δυνατόν πώς λειτουργήσαν οι διάφορε δράσει τα προγράμματα, ή πρωτοβουλίε, ώστε επιλεκτικώ να παραμένουμε στα καλύτερα. Υπό αυτήν την έννοια ανοίγει και η συζήτηση για τις αρνητικές προτεραιότητες, δηλαδή ενδεχομένως αναδιοργάνωση της ιεράρχησής μας. Μπορεί στο παρελθόν να είχαμε ακολουθήσει κάποιες ε, προτεραιότητες που δεν ήταν αναγκαστικά λανθασμένες, αλλά για λόγους ιστορικούς, λόγω των συγκεκριμένων συγκυριών, έχουν γίνει πλέον παροχημένες. Άρα ανοίγει πάλι η συζήτηση, ιδίως... Ε, μια συζήτηση που θα πρέπει να συνδεθεί με τα όσα λέμε στην Επιτροπή των Προλογισμών. Το να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας σε προτεραιότητες συγκεκριμένες, ε, ισχυρές και ε, πολύ σαφείς σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και τη διασπάθηση των κονδυλίων. Κάτι που βεβαίως θα μας οδηγήσει να σχεδιάσουμε έναν αποτελεσματικό προπολογισμό. Θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Ε, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η απόφαση να ε, προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων, γιατί νομίζω ότι ε, τώρα πλέον γνωρίζουμε όλοι μας καλύτερα πώς σκεφτόμετα, μπορούμε να προετοιμάσουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Και κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι βλάπτει μέσα από μια αποτελεσματική συζήτηση να εκμεταλλευτεί κανεί καλύτερα το χρόνο για να καταλήξει σε καλύτερε αποφάσει. Ε, νομίζω καλά τα κάναμε μέχρι τώρα ε, και ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε επικοδομητική συνεργασία. Σα ευχαριστώ. Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt aufrufen. Wir kommen damit, wie besprochen und im Programm verändert, zu der Debatte über den. Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση για το σχέδιο έκθεσης της ενδιάμεσης αξιολόγησης του ερευνητικού προγράμματος εδώ έχουμε εισηγητή τον κύριο Οντί. Ο κύριος Οντί θα ε, μιλήσει τώρα και μετά βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσία της εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους ε, εκπροσώπους του Συμβουλίου. Βοήθησαν πολύ στην προετοιμασία του θέματος στην αξιολόγηση πιο πολύ, όχι στην αναθεώρηση. Λοιπόν, θα σας πω ποιο είναι το πλαίσιο της έκθεσης αυτής. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο το ψηφίσαμε το 2006. Αποτελεί ένα στοιχείο της αναθεώρησης της στρατηγικής της Λισαβόνας που είχε ως στόχο, θα το θυμόσαστε όλοι, να κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον χώρο της γνώσης τον πιο ανταγωνιστικό στον κόσμο το 2010. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με 53-54 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια. Να το συγκρίνουμε με τα 17 του έκτου προγράμματος πλησίου. Πριν ήταν 5 χρόνια, τώρα είναι 7 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει η διαφορά του ποσού είναι τεράστια. Η έκθεση που σας προτείνω εγώ δεν αναφέρεται παρά μόνο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. θεώρησα ότι έπρεπε να μιλήσουμε μόνο για το 7 Για ποιο λόγο. Γιατί από τότε που ξεκίνησαν οι πολιτικές ε, διαβουλεύσεις βασιστήκαμε στα εξή. Πρώτον, πρέπει ναι ή όχι πολιτικά να βασιστούμε στην ε, χρήση του προγράμματος αυτού. Δεύτερον, απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας και έτσι τώρα έχουμε την στρατηγική 2020 όπου η έρευνα ξανά αναφέρεται σαν στοιχείο ανταγωνιστικότητας για την εσωτερική μας αγορά και υπέρ της ε, ευημερία των πολιτών μας. Έπειτα, είχαμε με τις εκλογές ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτο, τρίτη αλλαγή, το πρόγραμμα πλαίσιο το διαπραγματευτήκαμε και το αποφασίσαμε το 2006, πριν από την κρίση. Τώρα είμαστε 2011, εν μέσω της κρίσης και έχουμε ακόμα 2011, 2012 και 2013, χρονιές ε, κατά τις οποίες θα βγούμε από την κρίση, πολύ εύθραυστες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς θα χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό εν μέσω αυτής της ε, έφραυστης κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια δαπανήθηκαν 26 δισεκατομμύρια από ό,τι φαίνεται σε τέσσερα χρόνια, άρα για τα τρία χρόνια που μένουν έχουμε 29. Προ... Και συνδεσμεύσεις με το πρόγραμμα είναι ότι το 2013 τα χρήματα θα δαπανηθούν και το 2014 και το 2015 κατά πάσα πιθανότητα, γιατί πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί και να ξεκινήσει το 8ο μετά έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα σχετικά με την αξιολόγηση. Πρώτα απ' όλα, ε, μπράβο, το παμε και χτες ε, στην παρουσίαση, ε, συγχαρητήρια για την αξιολόγηση των ανεξάρτητων αξιολογητών. Έχω όμως να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Επαναλαμβάνω ότι εμείς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχουμε μια σφαιρική άποψη για το τι γίνεται με την έρευνα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει, ε, ε, άλλες υπηρεσίες. Έπειτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια περιοχή, φυσικά, αλλά από την άλλη έχουμε και τα διαθροτικά ταμεία. Τα διαθροτικά μας ταμεία όμως έχουν λισαβονοποιηθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, λέει ο μιλήτης, και έτσι δεν έχουμε σφαιρική άποψη. Τρίτο στοιχείο. Και εδώ ρωτάω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είχαμε αξιολόγηση για το ειδικό πρόγραμμα για την ε, Ευρατόμ. Υπάρχει το κύριο πρόγραμμα στο οποίο αναφερόμαστε, αλλά υπάρχει και ένα ειδικό πρόγραμμα πάνω από 2 δισεκατομμύρια το οποίο ολοκληρώνεται το 2011 μάλιστα και έχει να κάνει με την Ευρατόμ. Δεν πήραμε όμως αξιολόγηση γι' αυτό, σε αντίθεση με αυτό που προβλέπει το κείμενο του ειδικού προγράμματος. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να το είχαμε και αυτό, γιατί βλέπετε σήμερα το απόγευμα θα συζητήσουμε για τα πυρηνικά. Και το πρόγραμμα αυτό είχε σαν στόχο την έρευνα για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία από τα πυρηνικά. Τέσσερις μήνες ε, χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας, κάνει την, ε, να μας δώσει την ανακοίνωση, ενώ εγώ μέσα σε τέσσερις μέρες ετοίμασα τη δυο μου έκθεση. Έρχομαι τώρα στην έκθεση αυτή καθ' αυτή. Παράγραφος 3. Ε, το έβδομο ε, πρόγραμμα πλαίσιο αποδεικνύει ή όχι επαρκή ευρωπαϊκή προστιθέμενη εξία. Εγώ λέω όχι. Παρ' όλα αυτά έχω έτοιμη μια τροπολογία για να πω ναι τι εννοώ όμως εδώ. Εννοώ ότι αυτή η προστιθέμενη αξία δεν είναι προφανής. Και κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι ότι επειδή είναι περίπλοκο το θέμα, οι διάφοροι φορεί θεωρούν ότι η προστιθέμενη αξία, κυρίω όσον αφορά την απλοποίηση, δεν έχει επιτευχθεί. Και δεύτερον, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά μέσα που μερικές φορές αναρωτιόμαστε οι διάφοροι ειδικοί μερικές φορές ζητάνε να σταματήσουμε. Γιατί καταλήγουμε να αναρωτιόμαστε τελικά υπάρχει πιλότος στο αεροπλάνο. Γι' αυτό ετοιμάζω μια τροπολογία για να αλλάξω την ε, παραγραφό αυτή. Έρχομαι τώρα στην συνεργασία. Φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο. Υπάρχει διάρθρωση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που επίσης είναι αναγκαία. Ε, διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνα. ναι, και έχω και μια παράγραφο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Ε, ήρθε η ώρα. Αν θέλουμε να έχουμε όντω πιλότο μέσα στο αεροπλάνο το Μάιο, πρέπει να αναρωτηθούμε. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να διαρθρώσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα για να λαμβάνει υπόψη και τα οικονομικά μέσα και τη στρατηγική και να έχει και μια πολιτική αυτονομία. Στην παράγραφο 14, από την άλλη, προτείνω μια τροπολογία για την άμυνα. Διότι έχουμε νομική βάση στη συνθήκη και σας προτείνω να συζητήσουμε. Μήπως ήρθε η ώρα να έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την βιομηχανία άμυνας. Θα υποβάλω τροπολογία πάντως ώστε η παράγραφος που έχει να κάνει με το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο να είναι χώρια, γιατί έτσι όπως διατυπώνεται εδώ είναι σαν να μην υπάρχει νομική βάση. Θα αποσύρω λοιπόν αυτή τη σύνδεση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά την παράγραφο θα την αφήσω για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Στην παράγραφο 17 τώρα προτείνω την εδαφική κατανομή των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης. Η ιδέα είναι να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία, που γίνεται τοπικά έρευνα και περιφερειακά, και να δούμε μήπως πέρα από τη χρηματοδότηση της αριστείας, μήπως μπορούμε να έχουμε και μια κατανομή των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περισσότερο θέμα τοποθέτησης της έρευνας αυτής, γιατί καλό είναι να ε, κατανέμεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παντού έχουμε επιστημονικές διάνοιες. Το θέμα είναι να υπάρχει μια συνοχή σε αυτά που γίνονται και προτείνω στην ατολική σκέψη, όχι στην έκθεση, να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες και κάποιους ε, τρόπους ώστε ε, να μπορούν μεταξύ τους να συνεργαστούν οι διάφοροι ερευνητές και να επικοινωνήσουν ε, μαζί τους, έστω και από μακριά, ώστε να ξέρουν ε, τι, ο ένας τι κάνει ο άλλος. Για τη χρηματοδότηση τώρα και την... και όλα όσα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος, επιμένω στην καινοτομία. Και έρχομαι τώρα και στην απλοποίηση. μέτρα απλοποίηση. Μην απομακρυνθούμε από την έκθεση Καρβάλιο. Εγώ άκουσα τον αξιολογητή χτες που αναφερόταν στον αποδεκτό ε, βαθμό κινδύνου. Αν το κάνουμε αυτό για την έρευνα πολιτικά, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο, ότι στην έρευνα δεχόμαστε να κάνουμε παραπάνω λάθη. Οι επιστήμονες να κάνουν επιστήμη και οι ελεγκτές να κάνουν έλεγχο αλλά να υπάρξει μια ομάδα εργασίας της δικιάς μας Επιτροπής και της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, ώστε στην μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού να μπορέσουμε πολιτικά να βάλουμε τις νομικές βάσεις που είναι αναγκαίες για να συμπεριληφθεί η έκθεση Καρβάλιο. Αυτό προτείνω εγώ. Και όχι να διακινδυνεύσουμε τίποτα. Αυτά είχα να πω Αγαπητοί συνάδελφοι, περιμένω τις αντιδράσεις σας. Έτσι κι αλλιώς θα προσπαθήσω με τους ε, σκιώδεις από διάφορες πολιτικές ομάδες να καταλήξουμε σε συμβιβασμού ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή υπεραξία, για τους στόχους απέναντι στη βιομηχανία και τέλος μήπως πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορούμε μέσα στα τρία επόμενα χρόνια για κάθε νέο πρόγραμμα να λάβουμε υπόψη μας τις μεγάλες ε, οι υποδομές που υπάρχουν ήδη για τα θέματα τα οποία εντόπισαν ε, οι ειδικοί, γύρανση του πληθυσμού, ενέργεια, κλίμα. Γιατί να μην βάλουμε και κάτι για τον καρκίνο. Να είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο. Βιοτεχνολογίες. Κάποια θέματα δηλαδή όπου εμείς Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο υπέρ της ευημερία των πολιτών μας και υπέρ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεν έβαλα το ρόλο των γυναικών. Περιμένω βέβαια πολλές ε, τροπολογίες πάνω σε αυτό. Αυτά κύριε Πρόεδρε είχα να πω. Καταλαβαίνω ότι είναι ατελής η έκθεσή μου. Ζητώ επίκαια γιατί είχα λίγο χρόνο στη διάθεσή μου να την ε, ετοιμάσω εγώ και οι συνεργάτες μου, τους οποίους και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να δώσω το λόγο ε, ως πρώτη στη συνάδελφο κυρία Τόμσον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ουντή για την πολύ καλή ε, δουλειά του όσον αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα του είδους του στον κόσμο και η αξιολόγηση θα είναι σημαντικό και για το υπάρχον πρόγραμμα αλλά και για το επόμενο στρατηγικό πλαίσιο. Νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα προσφέρει τις απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη τόσο αλλαγές στην κλιματική αλλαγή και στη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο Ευρώπη, με θέμα την Ευρώπη ως ανταγωνιστή θα ήθελα να αναφέρω κάποιες ε, προτεραιότητες που νομίζω ότι είναι σημαντικές για αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό η αναθεώρηση να εστιαστεί στο βασικό πρόβλημα του 7ου ε, προγράμματος πλαίσιο που είναι η γραφειοκρατία. Χρειαζόμαστε μια έκθεση για το 7ο πρόγραμμα που να αναφέρεται ότι η απλούστευση χρειάζεται τόσο στο πρόγραμμα πλαίσιο όσο και στα επόμενα. Και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ε, αναφέρεται στο σχέδιο του προγράμματος ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει απλούστευση. Ένα άλλο σημαντικό μάθημα από το 7ο πρόγραμμα είναι ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία κυρίως όσον αφορά ε, τα διάφορα κεφάλαια. Χρειαζόμαστε μια ευέλικτη προσέγγιση που θα διασφαλίζει ότι μπορούμε να εκταμιεύουμε χρήματα όπου γίνεται έρευνα. Ε, τα άκαμπτα, ε, οι άκαμπτες δομές δεν πρέπει να αποτελούν φραγμό για την έρευνα. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δεν αναφέρονται επαρκώς στο σχέδιο της έκθεσης και όταν ήμασταν εδώ και τροποποιήσαμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου υπογραμμίσαμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ε, διακλαδικότητα και με τη δομή που έχει συσταθεί δεν βλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα διακλαδικότητας. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να μπορεί κανείς να συνδυάσει διάφορους τομείς της έρευνας. Επίσης ε, θα ήθελα ε, να μιλήσω λιγάκι για τη γνώση. Νομίζω είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι είναι απαραίτητο να συνδοθεί η έρευνα με την ε, παιδεία και τη βιομηχανία. Και έτσι θα έχουμε πολύ καλή γνώση. Όταν μιλάμε για τη βιομηχανία νομίζω πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Βλέποντας τις άλλες εκθέσεις, εκεί γίνεται λόγος για τη βιομηχανία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά τι είδους βιομηχανία και τι είδους ΜΜΕ, γιατί ε, δεν είναι όλες οι μικρομεσαίες στην Ευρώπη έτοιμες να συμμετάσχουν στα ερευνητικά προγράμματα. Θα ήθελα επίσης ε, να γνωρίζω, όταν μιλάμε για μεγάλες ε, βιομηχανίες, τι είδου δυνατότητες υπάρχουν να συμμετέχει και για να συμμετέχουν οι θαλάσσιες μεταφορές, ε, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές ε, σε πολλά κράτη-μέλη. Το επόμενο θέμα είναι η διάσταση του φύλου. Γνωρίζουμε ότι το 64% των ε, πανεπιστημίων στην Ευρώπη σήμερα είναι γυναίκες και ο στόχος μας είναι 40% συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ε, μάλλον το 64 ήταν άντρες, τώρα είναι 24 είναι γυναίκες και στόχος είναι το 40%. Εγώ είμαι συντονίστρια στην Επιτροπή Γυναικών και έχουμε καταρτήσει κάποιες προτάσεις για αυτή την έκθεση και τις ψηφίσαμε στην Επιτροπή Γυναικών με απόλυτη ομοφωνία. Έτσι λοιπόν εξετάζουμε και το θέμα του, α, ε, της ποσότητας των γυναικών Χτες ε, είπα, αλλά και σήμερα θα επαναλάβω, το θέμα της αριστείας και το να ε, διασφαλίσουμε την αριστεία για όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει τις ε, υποδομές έρευνας ε, εκεί που δεν υπάρχουν και να ε, προάγουμε την έρευνα μέσα από τα περιφερειακά ταμεία. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στα κρατημέλη, επιστημονική πολιτική των κρατών μελών, στην έρευνα γενικότερα να υπάρχει καλύτερο συντονισμός και θεωρώ ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ ε, με αυτά που ελέγχθησαν χτες. Ε, πράγματι το πρόγραμμα αυτό είχε ε, θετικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή υπεραξία. Προσβλέπω ε, σε περαιτέρω συνεργασία για το πρόγραμμα αυτό, σε συνεργασία με τον κύριο Οντί και τους άλλους σκιώδης συγητές. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα όπως ο συνάδελφος να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Ντί για την δουλειά του. Να πω απευθείας ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις που μας έχει υποβάλει. Μου φαίνεται προφανές ότι εδώ πρέπει να υπάρχει και υπάρχει συνέχεια μεταξύ της έκθεσης που μας υπέβαλε η κυρία Γκράσα Καρβάλιου και ε, των όσων εδώ ανακτώνται κατά κάποιο τρόπο στα πλαίσια του εβδόμου προγράμματο προγράμματος πλαισίου. Ε, επίσης μας ενδιαφέρει και ποια είναι η γενικότερη κατεύθυνση του Κοινοβουλίου για τις εκθέσεις που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία και τον ορισμό των προγραμμάτων πλαισίων. Δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις διότι νομίζω ότι θα έχουμε δυνατότητες να συζητήσουμε με λεπτομέρειες όλα αυτά τα θέματα. Κάποια σύντομες παρατηρήσεις απλώς σε σχέση με την έκθεση που μας υποβλήθη. Σημερίζομαι πολλές από τις παρατηρήσεις που γίνονται, ιδίως ό,τι φορά τη διάσταση των ανθρώπων που ξέρουμε ότι συμμετέχουν σήμερα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όμως, σε σχέση με αυτά πρέπει να πω ότι νομίζω θα έπρεπε να έχουμε την τόλμη να πάμε ακόμη πιο μακριά σε σχέση με τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε, διότι ήδη αντοπίσαμε κάποια θετικά στοιχεία από την αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου, οπότε... Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς όπου έγιναν συγκεκριμένες ε, παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε στου τομείς αυτής εργάζονται άνθρωποι. Να κοιτάξουμε λοιπόν την κινητικότητά τους, το ποιο, πώς υποφελούνται ή εξαρτώνται από τις υποτροφίες Marie Διότι η κινητικότητα δεν σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχει προώθηση της επιστημονικής σταδιοδρομίας του ερευνητή. Να Σκεφτούμε λοιπόν αυτό ως θέμα, την ανάγκη πρόθεσης της σταδιοδρομίας, ε, ανέλυξης επιστημονικής των ερευνητών, κάτι που αφορά πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επιπλέον, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε δύο στοιχεία που ανέφερε η προηγούμενη ε, συνάδελφος, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων και των γυναικών. Αυτή η ισορροπία και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να αναζητηθεί. Σε ένα άλλο σημείο της έκθεσης και το βλέπουμε ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, είναι αυτά που αναφέρονται στο 30. Δηλαδή, ανάγκη να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας. Εδώ βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Όπως σωστά αναφέρθηκε στην εκθεσή σας, μας μένουν ακόμη δύο χρόνια για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλαίσιο, οπότε θα πρέπει ένα μέρος της χρηματοδότησης να αποδοθεί στην αντιμετώπιση των αναγκών που δημιούργησε ακριβώς αυτή η οικονομική και κοινωνική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό λοιπόν θέτει και ένα νέο ερώτημα. Προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές. Προφανώς πρέπει να οριστούν από πολιτικής άποψης. Όμως πουθενά δεν γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Οι πολιτικές αυτές προτεραιότητες επέτυχαν τους στόχους τους ή όχι. Εδώ λοιπόν διαφωνώ με το σημείο 14. Ενίσχυει το τομέα της ασφάλειας. Είδαμε τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε δεδομένα αν χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Έχουμε εντοπίσει τα θετικά στοιχεία που μας αποδεικνύουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι προφανώς με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχαμε στη συζήτηση τη όλη αυτή τη έκθεση μέσω τη διαδικασία τροπολογιών και των συμβαστικών τροπολογιών, όμω θέλω να κάνω μια τελική παρατήρηση. Μου φαίνεται ότι το εργαλείο αυτό είναι τέτοια σημασία και η έκθεση αυτή τέτοιου βάρου και τέτοια βαρύτητα, που θα πρέπει να τα δούμε όχι μόνο ως στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφορών περιφερειών του κόσμου ω προ την έρευνα και την καινοτομία, αλλά για να εξασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή. Έχουμε ακόμη πολλέ ανισότητε μεταξύ των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλύτερη διάρθρωση του προγράμματος αυτού με τις ε, επιμέρους ε, πρωτοβουλίες εθνικές και περιφερειακές. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντί για την τόσο πλήρη έκθεσή του, η οποία αντάσσεται πάρα πολύ καλά στην σημερινή οικονομική κατάσταση. Δείχνει πώς πάει η στρατηγική μας όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα της συνέχισης της διαδικασίας απλούσταυσης που ξεκίνησε το 2010 και της μείωσης των διοικητικών φραγμών που έχουν σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η πρόσβαση πολλών στους διαγωνισμούς. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανακοίνωσή της για την απλούστευση είναι ενδιαφέρουσα γιατί μιλάει για καινούργιες λύσεις όσον αφορά την έρευνα και νέα οικονομικά μέσα. Χρειάζεται ανταλλαγή ε, πληροφοριών και απόψεων σίγουρα με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Είπαμε ξεκάθαρα ότι η εκπροσώπηση δεν είναι επαρκής, η συμμετοχή δηλαδή ορισμένων χωρών μελών όπως για παράδειγμα των νέων χωρών μελών. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, η ανακοίνωση του Συμβουλίου λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει έκθεση για την ανεπαρκή αυτή αντιπροσωπευτικότητα και να προτείνει λύσεις για να διορθωθεί η κατάσταση και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλη. Ε, ε, πρόεδρε, ευχαριστώ να συγχαρώ και εγώ την, τον εισηγητή μας τον κύριο Ντέ για την εξαιρετική του έκθεση. Απλώς θέλω να προσθέσω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις που λόγω έλλειψη χώρου στο έγγραφο ε, ο κύριος Οντή δεν μπορούσε να τα συμπεριλάβει. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ό,τι χρήζει αλλαγής. Στις θεματικές προτεραιότητες έχουν προκύψει νέες που δεν υπήρχαν όταν σχεδιάστηκε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ενέργεια. Έμφαση στο ρόλο των ευρωπαϊκών φορέων στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, στην ενέργεια, ενώ για τη δομή. Για τη δομή να πω ότι πρέπει οι συνεργασίε στην έρευνα και τα σχετικά μέτρα να παραμένουν στο επίκεντρο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Επίσης, το μέρος που αφορά τις μεγάλες αλλαγές. Όμως, ακόμα και στο τμήμα που αφορά την συνεργασία, τα στοιχεία τη συνεργασία, πρέπει να προβλέψουμε κάποια προσαρμογή, συνδυασμό της προσέγγισης bottom-up, με μια περισσότερο πολιτικό στοχοθετημένη ατζέντα. Έτσι, τα όσα γίνονται τώρα για τα ICT και τις νεοαναδιόμενες τεχνολογίες μπορούμε να τα συναρμόσουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε εδώ και νέες ιδέες στα πλαίσια των προγραμμάτων συνεργασίας. διότι προφανώς θα προκύψουν νέες τεχνολογικές εξελίξεις στα πλαίσια του ICT. Εδώ τώρα για τις υποδομές. Το σύστημα των υποτροφιών Marie Curie έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει να προωθηθεί και για τις κοινέ τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βοηθηθούν με δικές μας προσαρμογές. Πρέπει αυτές οι πρωτοβουλίες να ανοίξουν στη συμμετοχή των μικρομεσαίων και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν από προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για αυτές. Και επίσης θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και ένα εργαλείο για την κατάλληλη αποτίμηση των αποτελεσμάτων, όπως προκύπτουν από την εκτέλεση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή νέων επιστημόνων όχι μόνο των ανθρώπων που αναφέρατε, αλλά και σε επίπεδο συνεργασία τα ερευνητικά προγράμματα μπορεί να σχεδιαστούν έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και να συμμετέχουν νεότεροι ερευνητές για την απλούστευση. Συμφωνώ απολύτω με την προσέγγιση του κυρίου ότι πρέπει να δούμε την έκθεση της απλούστευσης και να την αξιοποιήσουμε για να κάνουμε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο όλα όλα όσα δεν έκανε η Επιτροπή και ακόμη προλαβαίνουν να γίνουν. Χωρίς αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια ώστε στην ενδιάμεση αναθεώρηση να μπορούν να γίνουν αμέσως κάποια πράγματα χωρίς παρέμβαση της Επιτροπής. Η κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντί παρουσίασε πράγματι ένα έγγραφο πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλά δομημένο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά θα ξεκινήσω από το ίδιο που είπα και στην Επίτροπο εκείνη σήμερα το πρωί. Δηλαδή μια τέτοια αξιολόγηση 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει δύο συνέπειες. Η μία είναι μεσοπρόθεσμα Δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα εντοπίστηκαν ως καλά ή ως λιγότερο καλά και να χρησιμεύσουν για το σχεδιασμό του επόμενου προγράμματος, του 8ου προγράμματος πλαισίου. Δεν μπορούν να βοηθήσουν μερικά πράγματα τώρα μέσω για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Τη στιγμή που έχουμε ήδη γκρίνει πράγματα για το 2012 και μετά αλλά να δούμε και τι νομοθετική αναθεώρηση χρειάζεται ενδεχομένως. Η δεύτερη, εν πάση περιπτώσει, συνέπεια είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν ακόμα να αλλάξουν και να τεθούν σε εφαρμογή στο πρόγραμμα το σημερινό, το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο που πάει μέχρι το 2013. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω εδώ, βάσει μιας πρότασης του κύριου Οντί, που πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για την παράγραφο 14, όπου η έκθεσή του λέει κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και το ανέφερε και αυτός εξάλλου. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμεύσει ακόμα για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αναφέρομαι λοιπόν στην παράγραφο 14 στον τομέα της τεχνολογίας άμυνας. Η πρότασή του είναι πολύ σημαντική. Δεν βλέπω βέβαια να γίνεται τώρα τα δύο επόμενα χρόνια. Βλέπω όμως να γίνεται στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Όμως θα μπορούσε να γίνει τώρα το εξή στο θέμα των τεχνολογιών διπλής χρήσης με επιπλέον πόρους γίνεται να αναπτυχθεί η προπτική αυτή πιο απλά και πιο χρήσιμα τώρα για το υπόλοιπο του 7ου προγράμματος πλαισίου. Και θα έπρεπε το ίδιο να το κάνουμε και για άλλα πράγματα, για την ε, αδειοδότηση, όπου μπορούμε την αξιολόγηση να τη χρησιμοποιήσουμε τώρα. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα και στην αρχή, ότι η αξιολόγηση χρησιμεύει αφενός για να ε, σχεδιάσουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, αφετέρου για να βελτιώσουμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο στο χρόνο που του μένει. Έρχομαι τώρα και στην παράγραφο 17, όπου προτείνεται η εδαφική κατανομή των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου, εδώ λοχεύουν κίνδυνοι. Υπάρχει μια αντίφαση δηλαδή. Αν δούμε τόσα έχουμε πει για την αριστεία και τις πολιτικές έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο πράγμα είναι τους πόρους να τους κατανέμουμε εδαφικά, των διευθυντικών ταμείων δηλαδή, και άλλο είναι αυτό. Γιατί με τέτοιου είδους διατυπώσεις υπάρχει κίνδυνος. Επειδή θέλουμε να πετύχουμε μια εδαφική κατανομή, τελικά παραβιάζουμε τις αρχές που διέπουν την έρευνα. Και για να πετύχουμε κάτι που να ικανοποιεί τους πάντες, χάνει τη φύση της η αρχική μας βάση για την έρευνα. Η έρευνα χρειάζεται απλούστευση, χρειάζεται ελαστικότητα στη διαχείριση, χρειάζεται οικονομικά μέσα, τα κατάλληλα και όλα αυτά για την εξυπηρέτηση της έρευνας που βασίζεται στην αριστεία. Τα υπόλοιπα μπορούν να ταχατοποιηθούν με κατανομή των πόρων κλπ. Αλλά προσοχή, μην πλήξουμε την ε, έρευνα με τη διατύπωση αυτή περί εδαφικής κατανομής. Ευχαριστούμε, ο κύριο Ευχαριστώ τον κύριο Ντί. Όντως, ε, ε, σημειώνει εδώ ότι πρέπει να συζητήσουμε συζητήσουμε ακόμα. Εγώ θέλω να έρθω στο θέμα της ε, πρόσθετης αξίας στην οποία αναφέρθηκε ο ίδιος ο Αυτό είναι το κλειδί των συζητήσεων μας, γιατί είναι εύκολο να πούμε προσθεθέμενη αξία. Μερικές φορές μας φτάνει να προσθέτουμε πόρους σε αυτά που δίνουν τα κράτη-μέλη, οι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Και τότε λέμε ότι έχουμε προσθεθεμένη αξία. Εγώ ομως δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ νομίζω ότι η προσθεθέμενη αξία πρέπει να είναι η αριστεία που μπορούμε να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να συνεισφέρουμε στην δημιουργία δυναμισμού, να δημιουργήσουμε αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περί αυτού πρόκειται. Τότε ε, μιλάμε για προστιθέμενη αξία και αυτό πρέπει να κάνουν τα προγράμματα πλαίσιο. Δεν φτάνει η επένδυση. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό που πολλές φορές προσπαθούν να κάνουν τα κράτη-μέλη από μόνα τους. Γι' αυτό και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για ενταφική κατανομή. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα συζητάμε ίσως στα πλαίσια της συνεργασίας ή των διαφορετικών ταμείων. Αλλά προστιθέμενη αξία μπορούμε να έχουμε στην έρευνα μόνο αν πετυχαίνουμε αριστεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πολλά έχουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, μεγάλες ε, επενδύσεις για την έρευνα. Αυτές θα είναι εφικτές μόνο εφόσον υπάρχει συνεργασία. Το κόστος, οι επενδύσεις είναι τόσο τεράστια που τα κράτη-μέλη από μόνα τους αποκλείεται να επενδύσουν και να μπορέσουν να υποφεληθούν από μια τέτοια επένδυση αν η επένδυση αυτή δεν γίνεται από κοινού. Έπειτα, το Marie Curie που έχει να κάνει με την κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι για να δημιουργηθεί αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος ε, επιστήμης. Πρέπει όμως να χρησιμοποιηθούν όλοι οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτυχία. Και έτσι δίνουμε απαντήσεις και στις ανησυχίες υπέρ των νέων ερευνητών ή των γυναικών ε, ερευνητριών. Χρειάζεται κινητικότητα να πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν ευκαιρίες. Αυτόν τον χαρακτήρα κινητικότητας θα ήθελα να τον ενισχύσουμε, να προσθέσουμε κάτι σαν ένα βάουτσερ για την έρευνα ή να βρούμε κάτι άλλο. Να μην υπάρχει μόνο η χρηματοδότηση, να υπάρχει για την έρευνα, αλλά να υπάρχει και ε, η σωστή διάνοια που θα πηγαίνει εκεί κάθε φορά. Τέλος, το θέμα της πιστοποίησης πάντα επιστρέφουμε σε αυτό και σωστά. Όταν συναντιέστε με ανθρώπους στα πανεπιστήμια ή στις επιχειρήσεις, αυτό πάντα αναφέρουν. Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα από ό,τι ήταν ε, στα προηγούμενα προγράμματα πλαίσιο, αλλά εξακολουθούν να μένουν πολλά να γίνουν. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί μπορεί να ακούγεται σαρκαστικό, αλλά μερικές φορές έχουμε την τάση να κοιτάμε τα πανεπιστήμια που υπάρχουν 500 χρόνια τώρα, 100 χρόνια και τα βλέπουμε σαν ύποπτα ιδρύματα που θα κάνουν καταχρήσεις, θα πάρουν τα λεφτά και θα φύγουν. Δεν λέω για τη χώρα μου. Αλλά να για παράδειγμα την Σορβόνη. Αν πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να τα. Το ίδιο ισχύει και για τη Χαδεβέρ, για τη Σαλαμάνκα, Πολώνη. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να αρχίσω να παριθμίζω πανεπιστήμια. Με την απλούστευση θέλαμε να πάμε πιο μακριά ακόμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαξίτης, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί πραγματικά συνέταξε ένα πολύ καλό έγγραφο και το ε, έγγραφο αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συζητηθεί και με βάση άλλους στόχους ε, της στρατηγικής 2020. Ε, ελέγχθησαν πάρα πολλά, δεν θέλω να το επαναλάβω, απλά θέλω να πω ότι στηρίζω αυτά που ελέγχθησαν ε, σχετικά με την απλούστευση ε, διοικητικών μέτρων. Αν δεν το πετύχουμε αυτό τώρα, τότε οι πράξεις μας θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτά που λέμε. Επίσης, νομίζω πρέπει να ορίσουμε με ακρίβεια τη δυνατότητα των ΜΜΕ, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να συμμετάσχουν στην έρευνα. Δεν έχουν ε, μεγάλες ε, δυνατότητες, ούτε πάρα πολλούς οικονομικούς πόρους, όμως ε, πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες πλαίσιο έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να συμβάλλουν στην υπεραξία στην Ευρώπη. Μιλάμε για δύσκολες ε, χρηματοδοτικές δομές που θα υπάρχουν στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να ε, εξελίξουμε τα μέσα και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Και όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή στην έρευνα, ο εισηγητής μίλησε για την εδαφική αρχή που θα ισχύει στο μέλλον. Και αυτό ε, θα είναι τουλάχιστον το ίμιση της λύσης, γιατί μερικές φορές μοιάζει να χάνεται ένα μεγάλο δυναμικό που υπάρχει στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να προσέξουμε καλύτερα το θέμα αυτό. Πρέπει επίσης να αποδώσουμε μεγαλύτερη σημασία και στη συμμετοχή νέων επιστημόνων. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον εισηγητή. Η έκθεση είναι ισορροπημένη και θα είναι χρήσιμη για όλους μας στο μέλλον. Λοιπόν, ε, τρεις ε, ε, θα έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, να είστε όμως σύντομοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλοι. Ο κύριος Βίμπα έχει το λόγο. Ναι, δεν θέλω να επαναλάβω όσα τόσο ωραία είπαν οι προλαλήσατες. Θέλω όμως να συγχαρώ παρόλα αυτά τον κύριο Ντί για την εκθεσή του. Εκτίμησε όλος ιδιαίτερος το γεγονός ότι δεν αποφεύγει το πρόβλημα της οργάνωση της έρευνας γιατί να μιλάμε για την απλούστευση κατά της γραφειοκρατίας δηλαδή, ναι. Αλλά αν θέλουμε να μην παραμείνουμε στα λόγια, αλλά να προχωρήσουμε και στην πράξη, πρέπει να προτείνουμε νέα δομή, νέα οργάνωση της έρευνας. Κατά τη γνώμη μου πάντως η αλλαγή του καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είναι πολύ σημαντικό, γιατί ζούμε ένα παράδοξο η έρευνα στις ευρωπαϊκές χώρες καθυστερεί. Δεν έχουμε πετύχει ούτε τους στόχους της Λισαβόνας, του 3% του προπολογισμού, είμαστε στο 1,8 ή 1,5, αλλά επιπλέον η καθυστέρηση και η απόστασή μας από τις ΗΠΑ και την Ασία μεγαλώνει. Και παρόλα αυτά δεν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον προπολογισμό που έχουμε εμείς ήδη προβλέψει. Τον έχουμε χρησιμοποιήσει στο 45%. Μας μένουν 28 δισεκατομμύρια για τα επόμενα τρία χρόνια. Και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν έτσι όπως έχουν σήμερα οι διαδικασίες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί τι νόημα έχει. Υπάρχουν λοιπόν προτάσεις και πρέπει να τις εξετάσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μια που σήμερα πρόκειται για ένα καθαρά εκτελεστικό όργανο. Πρέπει να αποτελέσει ένα νομικό όργανο, ανεξάρτητο όπως πολύ σωστά ε, σημειώνει και η έκθεση του καθηγητή Μπίνη, στην οποία αναφέρθηκα και χθε. Αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας πρέπει να αποκτήσει ε, πραγματικές εξουσίες απόφασης και να είναι υπεύθυνο όχι μόνο για την ερευνητική στρατηγική, αλλά και για την διοικητική διαχείριση. Μόνο έτσι, πιστεύω, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της απλούστευσης και της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Οντί για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Να σταθώ σε τρία σημεία που θεωρώ ουσιαστικά. Πρώτα απ' όλα, απλούστευση, συντονισμός, έλεγχος, βέλτιστες πρακτικές, Νομίζω αυτά έχουν ήδη σχολιαστεί. Έπειτα τα ερευνητικά κέντρα πανεπιστήμια και εταιρείες, ε, ερευνητικά κέντρα πρέπει να συντονιστούν. Πρέπει να υπάρχει μια πορεία παράλληλη, κοινή, ώστε να υπάρξει τέλεια διοργάνωση για να μπορούν πλήρως να έχουν διάλογο και συζήτηση μεταξύ τους όλοι αυτοί οι φορείς. Και τρίτη σημαντική παρατήρηση Πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Το ποσό αυτό που ανέφερε στα 29 δις είναι ένας πακτολός χρημάτων εάν καταφέρουμε να τον καλύψουμε γιατί μιλάμε εδώ για κονδύλια που δεν θα χαριστούν. Θέλουμε να δοθούν για να λειτουργήσουν τα προγράμματα, να δώσουν καρπούς, να, δώσουν, να έχουν κάποιο μέλλον. Δεν χρειάζεται πλέον να εκφραζόμαστε μόνο μέσω διαγωνισμών, αλλά αξιοποίησης, ρεαλιστικής αξιοποίησης των προγραμμάτων. Αυτό είναι που πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχει βουνό για, χρημάτων για την ανάπτυξη των οικονομιών αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα και για τη συνοχή. Ιδάλλως η έρευνα παραμένει ένα στοιχείο εθέριο. Δεν είναι πραγματικό. Εδώ θέλουμε κάτι πιο πεζό, κάτι πιο προσγειωμένο. Να έχουμε δηλαδή business για τις επιχειρήσεις. Ιδάλλως δεν έχει κανένα νόημα. Πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ στην ενδαφικοποίηση διότι είναι μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες που πρέπει να κάνουμε σήμερα προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, κύριε ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Σας άκουσα όλους. Και ξέρω ότι ο συνάδελφος δούλεψε με μεγάλη υπευθυνότητα και πολύ καλά. Ξέρω ότι είχε λίγο χρόνο στη διάθεσή του να ετοιμάσει την έκθεση. Πάντως κάποια από τα σημεία στην έκθεσή του με απασχολούν ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να διατυπωθούν διαφορετικά. Πρώτον, Υπάρχουν κάποια μηνύματα που μας ήρθαν από τις ομάδες, όπως του καθηγητή που ήρθε εδώ χτες, και που λένε ότι πρέπει να αλλάξουν τα μέσα που χρησιμοποίησαμε στην προηγούμενη περίοδο. Και γιατί. Αν το σχέδιό μας είναι η καινοτομία, πρέπει να δούμε πώς λειτουργήσε μέχρι τώρα. Αν δούμε λοιπόν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και την αξιολόγηση, το κλασικό θέμα της έρευνας ε, και της συνεργασία πάει πολύ καλά. Γιατί? Γιατί βασίζεται σε μια παράδοση που ήδη υπάρχει. Γιατί η έρευνα είναι κάτι στο οποίο έχει συνηθίσει η επιστημονική κοινότητα. Το θέμα της γνώσης εξαρτάται από τις αγορές. Η λογική είναι τελείως διαφορετική. Μην μπερδεύουμε όμως την αγορά με κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα, αν δεν καταλάβουμε καλά τι είναι η καινοτομία, κινδυνεύουμε να δώσουμε λάθος λύσεις. Η καινοτομία είναι η πρώτη φορά που κάτι εμφανίζεται. Αυτό σημαίνει καινοτομία. Όχι τα πράγματα στα οποία είμαστε συνηθισμένοι. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, να δούμε η καινοτομία μέχρι σήμερα πώς λειτουργήσε. Και αυτό πριν φτιάξουμε νέα όργανα. Το θέμα τώρα τη εδαφική κατανομής. Δεν νομίζω ότι καλά το λέμε. Διότι το Συμβούλιο μπορεί να καταλάβει ότι πρόκειται για την κατανομή χρημάτων. Εγώ λοιπόν θα ήθελα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμφωνήσουμε ότι η αριστεία είναι μια προτεραιότητα να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα του 7ου προγράμματος πλησίου για να προωθήσουμε την αριστεία. Και εδώ έρχεται η ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το οποίο δεν αναπτύχθηκε αρκετά μέχρι τώρα είναι τα προγράμματα και εγώ προτείνω να απαιτήσουμε από τα κράτη-μέλη ή τέλο πάντων να τους ζητήσουμε η Ευρώπη, η οποία συνήθως δεν έδινε χρήματα για τον προγραμματισμό, τώρα να δίνει σε προγράμματα τα οποία όμως καλύπτουν κάποιες προϋποθέσεις και εφόσον τα πανεπιστήμια δίνουν ερευνητέ για τέτοιους, που, στόχους που είναι η κινητικότητα για παράδειγμα. Στο Στάνφορντ δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το πόσο παλιό πανεπιστήμιο είναι ούτε και στην ε, Ισπανία η αρχαιότητα ενός ερευνητή λαμβάνεται υπόψη. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας για την κινητικότητα, το μάστερ ή τις υποτροφίες, μπορούμε να καταλήξουμε στο γερμανικό ε, σύστημα που άπαξ και είναι καλό ένα πρόγραμμα, αυτό φτάνει, τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε ένα 5-7% στα προγράμματα αριστείας. Δηλαδή, ο παράγοντας αριστεία να είναι καθοριστικός. Και πώς. Εντάξει, να ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μας βοηθήσει έρευνα, να μας βοηθήσει στο να το καθορίσουμε αυτό. Το Συμβούλιο θέλει να ξοδέψουμε λιγότερα χρήματα. Ναι, αλλά οι ερευνητές θέλουν ευρωπαϊκά προγράμματα, να δουλέψουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν τα θέλουν για τα υπουργεία τους. Γι' αυτό και πρέπει να επιμείνουμε στην αριστεία αυτή. Και τέλος, υπήρξε κάποιο λάθος νομίζω στην επικοινωνία. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρώπη δεν ξέρει τι είναι το πρόγραμμα πλαίσιο. Και το Flexia να ξέρετε ότι δεν το ξέρει ο κόσμος. Χρειάζεται μια ανακοίνωση ισορροπημένη όπου να ξεκαθαρίζουμε ότι η βασική έρευνα θα διατηρηθεί και θα προστατευτεί γιατί αλλιώς να ξέρετε ότι πανικοβάλλεται η επιστημονική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Και για άλλη φορά συγχαρητήρια στο φίλο Οντί. Δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου, αν και η Επιτροπή θέλει, να πάρει το λόγο. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλο ένα λεπτό κύριο Σοντή στη συνέχεια. Εντάξει, συμφωνείτε να είσαστε Πολύ σύντομη, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ σύντομα να εστιάσω την προσοχή μου σε τρία θέματα. Το ένα αφορά στην ευρωπαϊκή υπεραξία που αναφέρθηκε ως βασική έννοια. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι αυτό συζητήθηκε τόσο στην έκθεση Άρενμπεργκ που παρουσιάστηκε χθε, όσο και ε, την εκ αξιολόγηση του έκτου ε, προγράμματος ε, πλαίσιο. Έγινε μια μελέτη από τον συνάδελφο από την Αυστρία ε, και εκεί προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε όλες τις, όλα τα στοιχεία του προβλήματος. Κατόπιν αναφέρθηκαν αρκετά επιχειρήματα υπέρ της ευρωπαϊκής υπεραξίας των προγραμμάτων πλαίσιο. Ένα άλλο θέμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι ένα ερώτημα του κυρίου Οντί για το τι ακριβώς συνέβη με την ενδιάμεση εξολόγηση της Eurotom. Και να σας πω ότι από τότε που λειτουργεί το πρόγραμμα Eurotom σε διαφορετική νομική βάση και με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, ε, που κατ' ουσίαν προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί ε, το 2011 για το 2014. Γι' αυτό η αξιολόγηση του προγράμματος EuroTOM ε, έγινε πιο γρήγορα, ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2010 και η ενδιάμεση αξιολόγηση έγινε από τον πρόεδρο κύριο Μιλ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ε, Ομοσπονδίας Βιομηχάνων της Τσεχίας. Και το τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω είναι το τι ακριβώς κάνει η Κομισιόν όσον αφορά στα πορίσματα της έκθεσης Άρεμπακ. Θέλω να σας πω ότι στην ανακοίνωση αναφέρουμε μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες διεξάγονται αυτή τη στιγμή. Η μία ε, προφανώς έχει άμεση σχέση με το θέμα της απλούστευσης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Το δεύτερο έχει σχέση με τη διεθνή συνεργασία, ε, σημαντική αναθεώρηση του πώς πρέπει να προβληθούν τα βασικά στοιχεία σε αυτόν τον τομέα και το τέταρτο είναι ε, οι μετρήσεις, ε, η επόμενη θα γίνει τον Ιούλιο. Ε, θα αποδείτε μεγαλύτερη σημασία στι μεγάλες προκλήσεις και μεγαλύτερος προσανατολισμός για τον καθορισμό της στρατηγικής του 2020, πρωτοβουλία μιλωματική και κύριε Οντί, σας παρακαλώ τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, το εκρεμές δεν λειτουργεί σωστά. Είχα δύο λεπτά στη διάθεσή μου από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα ήθελα το ένα να το δώσω στο Συμβούλιο για να μας πει και εκείνο την άποψή του, αν μπορεί. Μήπως θέλει κανείς να πει κάτι από το Συμβούλιο. Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Ε, δεν είναι δυνατόν τώρα. Τι κρίμα. Γράψτε το στα πρακτικά. Λυπάμαι ιδιαίτερος, διότι είναι εξαιρετική η συμβουλή μας εδώ και δεν έχουμε καμία τοποθέτηση από τα κάτι μελη και το Συμβούλιο. θα είμαι πολύ σύντομο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για τι ευχαριστίε του και τα καλά του λόγια. Η έκθεση νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο είναι πραγματικά ακόμα μη πλήρη, αλλά θα λάβω υπόψη όλε τι παρατηρήσει που έγιναν, ιδίω για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, την εδαφική κατανομή. Η Πιλάρ ίσως να μην με άκουσε, αλλά νομίζω ότι είπα για τα νομικά μέσα του 7ου προγράμματο και τη σχέση έρευνα με άμυνα. Θα την διορθώσουμε αυτή την ασυνέπεια. Και για την εδαφική κατανομή. Να επιμείνω απλώ σε κάτι εδώ. Πόρο απέχω από την ιδέα να αφαιρέσουμε τη διάσταση της αριστείας από τους μεγάλους μου στόχους. Όχι, θέλουμε απλώς χρηματοδότηση για τις μεγάλες ευρωπαϊκές υποδομές, διεθνείς υποδομές. Εγώ θέλω την αριστεία και υπ' αυτήν την έννοια οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, οι τηλεσυνεδριάσεις, προκειμένου να ευωδοθεί η αριστεία, να προωθηθεί η εδαφική κατανομή. Όλα αυτά θέλουμε να μας οδηγήσουν σε μια ευρωπαϊκή ενότητα ως προς την αριστεία των επιμέρους περιφερειών, γιατί έχουμε πραγματικά επιστημονικές δυνατότητες παντού. Θα λάβω λοιπόν υπόψη όλες αυτές τι παρατηρήσεις και θα δω με του εισηγητέ των διαφόρων πολιτικών ομάδων ποια είναι τα βασικότερα μηνύματα που πρέπει να τονιστούν. Όχι μόνο για να εξελιχθούν οι αμφισημίε, διότι και ο τίτλο τη έκθεσης θα μπορούσε να αλλάξει. Όχι η αναθεώρηση, διότι δεν θέλουμε εδώ να ε, ανοίξουμε συζήτηση για την αλλαγή του κανονισμού αλλά θέλουμε να απευθύνουμε μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε το πρόγραμμα εργασιών τη, να λάβει υπόψη και την αξιολόγηση που έγινε και τις εντυπώσεις και τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Στις 20 Μαρτίου έχουμε την προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους συμμετάσχοντες στη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε που μείνατε ως το τέλος. Äh, ε, να δούμε βέβαια ότι κάποιες φορές δεν είναι ευγενικό που μερικοί έρχονται στην αίθουσα, καταχράζονται το χρόνο ομιλίας και μετά αφαιρούν χρόνο ομιλίας από άλλους, φεύγοντας ξαφνικά. Τέλος πάντων, εδώ οι περισσότεροι σήμερα ακολούθησαν την αντίθετη στάση. Σας ευχαριστώ πολύ όλου. Θα το πούμε το απόγευμα.